Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας παρακαλούσα συνάδελφοι να αποχωρήσετε πιο ήσυχα. Παρακαλώ ησυχία. Μην γίνονται τόσες πολλές συζητήσεις στην Ολομέλεια. Παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα. Uh, Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ. Sorry. Sorry. Συγχαρητήρια στον κύριο Γκαλτιέρη και στον κύριο Μπροκ. Συγχαρητήρια. Καθίστε όμως παρακαλώ. Ή φύγετε, ή καθίστε ή φύγετε. Καλή τύχη, συγχαρητήρια και στους δύο. Po głosowaniu pierwszym punktem Λοιπόν, επόμενο σημείο που έχουμε να εξετάσουμε είναι η δήλωση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 24-25 Μαρτίου 2011. Θα προχωρήσουμε τώρα, θα πάμε στη συζήτηση. Θα ξεκινήσει από ο, τον Ένικο Γκιούρι, εκπρόσωπο τον Υπουργό που εκπροσωπεί την, ε, την Υπουργό που εκπροσωπεί την Ουγγρική Προεδρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη. καλώς ορίζω τη δυνατότητα να εμφανιστώ ενώπιόν σας πριν από την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ξέρετε πολύ καλά ότι θα είναι πάρα πολύ εντατική αυτή η συνεδρίαση λόγω των απρόβλεπτων γεγονότων των τελευταίων δύο εβδομάδων. Θα ήθελα καταρχάς να διατρέξω τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γνωρίζετε ότι θα υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία επίσημη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα το Γενικό Οικονομικό Πακέτο που ελπίζουμε να εθετηθεί από του αρχικού κρατών και κυβερνήσεων, η Λιβύη και η Νότια Γειτνίαση και η Ιαπωνία. Θα ξεκινήσω λοιπόν με την οικονομική, οικονομική πολιτική και τα οικονομικά και πολιτικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υφετήσει το πακέτο, ελπίζουμε, ούτω ώστε να ανταποκριθεί στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Επιτρέψτε μου να κατονομάσω τρία βασικά στοιχεία ε, της δέσμης μέτρων. Πρώτα απ' όλα, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την έγκριση των προτεραιοτήτων για την οικονομική ενοποίηση και τις διαθωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ξεκίνησε αρχές του έτους με την παρουσία σε πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής της εκτής εκθέσεως για την ανάπτυξη. Συμπεριλαμβάνει διάφορες στάσεις πολιτικής που απαιτούνται για να ενισχυθεί η ανάκαμψη, να βοηθήσουμε την Ευρώπη να διατηρήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και να πετύχουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2020. Η πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τώρα θα ολοκληρωθεί με την την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των προτεραιοτήτων για την οικονομική ενοποίηση και τι εθνικέ αλλαγέ σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προετοίμασε η ΕΚΟΦΗΝ και, και το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Λοιπόν, το θέμα τη εκθέσεω που ετοιμάστηκε από την Προεδρία ε, υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων την περασμένη Δευτέρα. Τα κράτη-μέλη ε, θα ακολουθήσουν γενικού προσανατολισμού εν την προετοιμασία του Συμφώνου Σταθερότητα και Συγκλήσεω των προγραμμάτων και των προγραμμάτων εθνική μεταρρύθμιση που θα υποβληθούν τον Απρίλιο. Το Συμβούλιο, βάσει τη αξιολογήσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προβεί στη δική του αξιολόγηση και θα δώσει προσανατολισμό στα κράτη-μέλη τον Ιούνιο, όταν θα πρέπει να ληφθούν σημαντικέ Μάλλον είναι ακόμα στην προετοιμασία σημαντικέ αποφάσει για τον προπολογισμό στα διάφορα κράτη-μέλη. Η Ουγγρική Προεδρία στοχεύει να τελειώσει το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο στην ώρα του πριν από τον Ιούνιο, το Συμβούλιο του Ιουνίου του 2011. Ε, θα πρέπει να ενισχυθεί και η οικονομική διακυβέρνηση. Αυτή είναι μια άλλη πτυχή και σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασιστικό ρόλο να διδραματίσει. Το Συμβούλιο ήδη έκανε σημαντική αλλαγή. Οι Υπουργοί Οικονομικών και Οικονομία συμφώνησαν με την γενική προσέγγιση του Συμβουλίου σχετικά με τι έξι νομοθετικέ Προτάσει για την ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό το επίτευγμα δίνει τη δυνατότητα στην Προεδρία να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο. Όπω γνωρίζετε το Συμβούλιο έχει προθεσμία από πλευρά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρέπει να τηρήσει την προθεσμία. Ιούνιο 2011 είναι η προθεσμία. Μέχρι τότε πρέπει να υπάρξει πολιτική συμφωνία επί του πακέτου. Τέσσερι από τι έξι προτάσει υπόκεινται στη δικασία συναποφάσεω. Ξέρουμε ότι η προθεσμία που επιβάλλεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν δεσμεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν είναι. Αλλά παίρνω, εκμεταλλεύουμε την επίσημη αυτή περίσταση να ζητήσουμε την εργασία του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο. Θα στείλει ένα εφησυχαστικό μήνυμα προ τι αγορέ, κάτι τέτοιο, και πιο σημαντικό προ του πολίτε μα, οι οποίοι περιμένουν από εμά να διαφυλάξουμε το ευρώ και την ευρωπαϊκή οικονομία μαζί με το ευρώ. Άρα έχουμε κοινή ευθύνη και εμεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Πρωθυπουργό μα Πρόκειται να συναντήσει τους ηγητές και τους συντονιστές που είναι υπεύθυνοι για αυτό το πακέτο και ελπίζω ότι θα έχουμε μια καρποφόρα συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Το τρίτο στοιχείο είναι η αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού σωμαία μέσω νέο φιλόδοξου ε, δοκιμασίας ε, Αντοχή, αν θέλετε. Έχουμε και το σύμφωνο για το ευρώ και πρέπει να επεκταθεί και στα κράτη-μέλη εκτό ευρωζώνης που θέλουν να μπουν στο ευρώ και θα ανακοινωθούν ενδεχομένω τα πρώτα εθνικά σχέδια δράσης για να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Πέμπτο στοιχείο είναι η ολοκλήρωση των εργασιών για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθερότητα και η ενίσχυση της Ευρω... του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αναμένεται ε, η συμφωνία της Υπουργικής Συνεδριάσεως ε, της Eurogroup που θα γίνει στις 21, Μαρ... έγινε στις 21 Μαρτίου και θα δοθούν ιδέουσες πληροφορίες ε, λαμβάνονται υπόψη μάλλον και οι απόψεις του Κοινοβουλίου. Το έκτο στοιχείο είναι η τροποποίηση της συνθήκης κάτι που ψηφίσαμε μέχρι τώρα και επίσημη υιοθέτηση της αποφάσεως που τροποποιεί τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με τη σύσταση του μελλοντικού συστήματος με το μηχανισμό σταθερότητας για τα κράτη-μέλη και ευχαριστώ τα, το Κοινοβούλιο για τη θετική ψηφοφορία και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά από την πλευρά σας. Όπω βλέπετε, έχει επιτευχθεί πραγματική πρόοδο για την καταπολέμηση τη κρίση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ολοκληρώσει αυτέ τι εργασίε και στην επόμενη σύνοδό του θα υθετήσει ένα γενικό πακέτο μέτρων για να ανταποκριθούμε στην κρίση μέσω χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δημιουργηθεί, θα προλιανθεί το έδαφο για ανάπτυξη βιώσιμη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Σα στραφώ τώρα προ την νότια πολιτική γειτονία και τη Λιβύη. Στι 10 Μαρτίου είχαμε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και 11 Μαρτίου συμπεράσματο του Συμβουλίου και το ψήφισμα του ΟΗΕ 1973 ε, και έχουν εκφραστεί έτσι ανησυχίες για την παρούσα κατάσταση στη Λιβύη και καταδικάζεται η συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ομή καταστολή, η βία καταστολή που διαπράττεται το καθεστώ κατά του λαού τη Λιβύη. Βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι η προστασία του άμαχου πληθυσμού, των πολιτών και υποστήριξη για τη δυνατότητα που θα έχουν οι Λίβοι να πραγματοποιήσουν τι προσδοκίε του για μια δημοκρατική κοινωνία. Ο συνταγματάρχη Καντάφη θα πρέπει να παραιτηθεί από την εξουσία αμέσω. Το καθεστώ του έχει χάσει την νομιμότητά του και δεν είναι πλέον ένας συνομιλητής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τι είδου δράσεις έχουν αναλυθεί από το Συμβούλιο σχετικά με αυτό. Πρώτα απ' όλα να αναφερώ τις κυρώσεις. Στις 28 του Φεβρουαρίου το Συμβούλιο θέτησε σε χρόνο ρεκόρ αποφάσεις που εκάλυπταν περιοριστικά μέτρα κατά του καθεστώτος. Στις 10 Μαρτίου περαιτέρω κυρώσεις προσετέθησαν. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιάς, απαγόρευση ταξιδίων, εμπάρκο για τα όπλα, ε, και όλα αυτά μπορεί να είναι γιατί θα πόσο χρησιμοποιηθούν για εσωτερική καταστολή. Ε, και αυτά ξεπερνούν τα μέτρα που είχαν επιβληθεί από το προηγούμενο ψήφισμα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και τρίτο στοιχείο, τρίτος γύρος κυρώσεων προβλέπεται. Βάσει τη εντολή που δόθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 21 Μαρτίου, το Συμβούλιο υιοθέτησε σήμερα μέσω τη γραπτή διαδικασία την πρόταση τη Ουγγρικής Προεδρίας να επεκτηθούν τα προεριστικά μέτρα και σε άλλους Λίβιους ε, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα και αυτές οι κυρώσεις συμπεριλαμβάνουν ήδη την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης. Αυτές οι κυρώσεις προσετέσαν το Συμβούλιο. Και εμεί θέσαμε και το θέμα τη ασφάλεια εφοδιασμού ενέργεια στο πρόγραμμα. Οι υπουργοί συζήτησαν μέρη την πολιτική κρίση, τη συνέπεια πολιτική κρίση, στην ενεργειακή αγορά, την ενεργειακό εφοδιασμό, ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια και συμφώνησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαρκή από θέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, όμω η συζήτηση εκ νέου τόνισε το πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη και την ανάγκη που υπάρχει για ακόμα ισχυρότερη κοινή ενεργειακή πολιτική συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπω είναι η ποικιλομορφία όσον αφορά τις, των διόδων εφοδιασμού σενάρια. Ικανοποιήθηκε, το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση μετά την απόφαση 1973 του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ και υπογράμμισε αποφασιστικότητα να συμβάλλει στην εφαρμογή αυτή τη αποφάσεω. Το Συμβούλιο επίση καλωσόρισε τη Σύνοδο Κορυφή των Παρισίων και θεώρησε ότι είναι σημαντική συνεισφορά αυτή για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Με διαφοροποιημένη προσέγγιση, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένα όλα μαζί να κινηθούν και με αποφασιστικότητα μαζί με όλου του διεθνεί εταίρου, κυρίω με τον Αραβικό Σύνδεσμο και άλλου φορεί τη περιοχή, ούτω ώστε να εφαρμοστούν πλήρως αυτές οι αποφάσεις. Το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη θα υποστηρίξουν τις δράσεις που προβλέπει από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων και το μάχο πληθυσμού και στου τομεί τη περιοχή που απειλούνται. Θα, θα εξακολουθούμε εμεί να δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλου αυτού που πλήττονται. Και βεβαίω θα πρέπει σε μεταγενέστερο στάδιο να βοηθήσουμε τη Λιβύη να οικοδομήσει ένα δημοκρατικό κράτο και να αναπτύξει το κράτο δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται ούτω ώστε να δώσει υποστήριξη και ανθρωπιστική βοήθεια κατόπιν αιτήματο τη υπηρεσία του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων και σύμφωνα με το συντονισμένο ρόλο που μπορεί να παίξει ο ΟΗΕ. Αυτέ οι δράσει σέβονται πλήρω κατευθείαν γραμμέ του ΟΗΕ για τη χρήση στρατιωτική άμυνα και πολιτική άμυνα. Ο ύπατο εκπρόσωπο ζητήθηκε να αναπτύξει περαιτέρω σχεδιασμό σύμφωνα με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη 11η Μαρτίου, υποστηρίζοντα την ανθρωπιστική βοήθεια, την προστασία των πολιτών και τι σχετικέ επιχειρήσει και μέσω θαλασσίων μέσων για την επίτευξη των στόχων. Τα πάντα πρέπει να γίνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό σε συνεργασία με τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ και άλλου. Η πρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ενώση επαφέ με τον Γενικό Γραμματέα του και χώρε τη περιοχή συμπεριλαμβανομένη τη Τινησία και τη Αιγύπτου και δηλώθηκε ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να δρομολογηθεί κατεπηγόντως ούτω ώστε να επιτραπεί περαιτέρω εξέταση του θέματος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλο τη εβδομάδας. Έτσι περαιτέρω τα κράτη-μέλη υπογράμμισαν εκ νέου την αλληλεγγύη τους όσον αφορά τα κράτη-μέλη εκείνα που πιο άμεσα ε, πλήττονται από μεταναστευτικέ ροέ και επανέλαβαν την ετοιμότητά του να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη ανάλογα με την εξέλιξη. Η Ουγγρική Προεδρία έθεσε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εσωτερικών και Δικαιοσύνη του Φεβρουαρίου, που έγινε 24-25 Φεβρουαρίου. Η κοινή επιχείρηση Ερμή ξεκίνησε στα πλαίσια του Frontex και συνέβαλαν διάφορα κράτη-μέλη ε, με πόρου. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τι συνέβη όσον αφορά την εκένωση Ήδη στις 23 Φεβρουαρίου η Προεδρία ενεργοποίησε μηχανισμό προστα... πολιτικής προστασίας για να προστατευτούν, να εκενωθούν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τη Λιβύη και αυτή η απόφαση υποστηρίχθηκε και από την ύπατη εκπρόσωπο. Εμπνευσμένη από την αρχή που καθορίζεται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ποια είναι η ευθύνη για την προστασία, η Ουγγρική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να συντονίζει τις προσπάθειες που διενεργούνται πιο συγκεκριμένα για τους πρόσφυγες και για τα θέματα των μετανάστευση. Υπό το φω αυτό, Υπουργό Εξωτερικών Γιάννου Μαρτούνι μαζί με, τον Επίτροπο, με την Επίτροπο Βάλστρομ επισκέφτονται τώρα την, Αίγυπ, την Αίγυπτο και τα κοινά σύνορα με τη Λιβύη. Ο Υπουργό Μάρτον πήγε στα σύνορα και μίλησε με τις τοπικές αρχές και στη δήλωσή του στα σύνορα είπε ότι χωρίς αεροπορικές επιδρομές θα μπορούσε να αποφευθεί μια φόρητη κατάσταση, είναι υποέλεγχο η κατάσταση, χάρη στις Αιγυπτιακές αρχές. Για τρεις μέρες δεν υπήρξε εκροή κόσμου, κάποιοι Λίβοι αποφάσισαν να επιστρέψουν, αλλά βεβαίως η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ασταθής και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα έχουμε περαιτέρω εκροές πληθυσμού ή όχι. Στις 3 Μαρτίου πήγα στα σύνορα της νησίας Λιβύης, συνοδεύοντας την Επίτροπο Γεωργίευα για να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί και ακόμα η κατάσταση ήταν πολύ κακή. Χιλιάδες άνθρωποι την ώρα έμπαιναν στην την νησία από αυτά τα σύνορα. Και η εκένωση ήταν το σημαντικότερο θέμα στις 3 Μαρτίου και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κράτη-μέλη να επαναπατρίσουν επίσης και πολίτες που δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως μεταναστές εργάτες. Όσον αφορά την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ο Ούγγρος πρεσβευτή στην Τρίπολη εκπροσωπού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εκεί, δεν θα αποχωρήσει και συντονίζει διπλωματικέ προσπάθειε, προξενικέ προσπάθειε εκ μέρου των κρατών μελών. Όσον αφορά την νότια γυτνίαση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην έκτακτη σύνοδό του στις 11 Μαρτίου δήλωσε ότι οι δημοκρατικές εξεγέρσεις επιφέρουν δραματικές αλλαγές στην νότια γειτονία. Οι δημιουργούνται νέες ελπίδες και δυνατότητες για να δημιουργηθεί ένα μέλλον βάσει δημοκρατίας, πλουραλισμού, κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής δυσκριοσύνη. Θα πρέπει να δηλωθεί ότι ε, δεν το πρόβλημα μόνο, δεν υπάρχει βία μόνο στη Λιβύη και στον Παχρέν και στην Ιεμένη έχουμε και άλλες βιοπραγίες και θα πρέπει να είναι σαφές ότι η βία δεν είναι αποδεκτή στην Ευρώπη. Οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το μέλλον τους ειρηνικά και δημοκρατικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει όλα τα βήματα προς δημοκρατική μεταρρύθμιση των πολιτικών συστημάτων που θα επιτρέψουν ευμάρια τελικά δημοκρατία, πιο ανάλογη κατανομή του πλούτου και καλύτερη οικονομική επίδοση. Οι χώρε τη περιοχή χρειάζονται οικονομική και τεχνική υποστήριξη για να βελτιωθεί ο έλεγχο των συνόρων και τα μέτρα που διευκολύνουν τον επαναπτωτισμό των μεταναστών στι χώρε καταγωγή. Θα του βοηθήσουμε σε αυτό. Το Συμβούλιο στη συνεργασία με του άλλου φορεί θα υποβάλει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη δυναμικού για τη διαχείριση του, των μεταναστευτικών ροών και της μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσόρισε την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑΣ ΕΚΟΣΟ που προτείνουν σύμπραξη για τη δημοκρατία για κοινή ευμάρεια στην Νότια Μεσόγειο βάσει διαφοροποιημένης προσεγγίσεως, βάσει κινήτρων που θα συνεπιφέρει όλα τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο ε, εκλήθη να εξετάσει εντάχει τις προτάσεις της ανακοινώσεως και κυρίως τους όρους υπό τους οποίους η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τους εταίρους θα διευρυθεί. Για να ολοκληρώσω την παρουσίαση των ιδεών, επί των οποίων χρειάζεται γρήγορη δράση, πρέπει να αυξήσουμε την οροφή για, την επιχειρήσει για τις, τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Επενδύσεων στις μεσογειακές χώρες που κάνουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις και το Κοινοβούλιο επ' αυτού θα διαδραματίσει ρόλο και βασίζομαι στη συνεργασία σας. Θα πρέπει να θετήσουμε την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επανεπονδύσει στα, ε, τα ποσά που έχουν απομείνει από πρώτερε επιχειρήσει και μάλιστα εμπλεκομένου πρέπει να δουν ποιου όρου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμηση και Επενδύσεων μπορεί να λειτουργεί στα πλαίσια τη Νότια Γυτνία και θα πρέπει να κάνουμε μια πρόταση όσον αφορά πανευρωμεσογειακή ε, προσέγγιση ε, για να αναπτυχθεί η περιοχή. Και τέλος, μέχρι τον Ιούνιο 2011 πρέπει να εγκριθεί ο κανονισμός που διευρύνει τις δυνατότητες που θα έχει η Frontex. Είναι εκ των νου κάνε, θα σταματήσω εδώ, δεν θα μιλήσω για την Ιαπωνία, γιατί έχουμε νέο σημείο επ' αυτού στην ημέση διάταξη. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Επειδή συνέβησαν πολλά, βλέπετε, και ήθελα το Κοινοβούλιο να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα ε, των ζητημάτων που συζητήθηκαν και όσων συμβαίνουν. Ευχαριστώ κυρία μου, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Γκέρι, αξιότιμα μέλη. Όπως είπα την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο θα δημιουργήσει η Ευρώπη στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης και 25ης Μαρτίου θα φέρει μια πραγματική αλλαγή στους όρου του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια θα είναι ένας ακρογωνιαίο λύθο όσον αφορά μια περικτική απόκριση προς την κρίση και θα σηματοδοτήσει την απαρχή της πλήρους του εφαρμογή με τη σύσταση ενός νέου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και ελπίζουμε μια Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, η οποία στέκεται σταθερά στα δυο τη πόδια και δεν προχωράει χωλένοντας η οικονομική πολιτική της χώρας μέλης θεωρείται πλέον ότι αφορά όλη, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλες τις χώρες. Για πρώτη φορά θα έχουμε τα εργαλεία τα οποία χρειαζόμαστε για μια πρώιμα και ισχυρό συντονισμό όλων των πολιτικών πριν κάθε χώρα μέλος ε, δημιουργήσει τη δική της πολιτική και καταρτήσει το δικό της προϋπολογισμό για το επόμενο χρόνο. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε μαζί με την ε, οικονομική πολιτική και την πολιτική του προϋπολογισμού ταυτόχρονα. Ε, θα έχουμε η ετήσια μελέτη παρουσιάζει 10 προτεραιότητες οι οποίες όλες ε, εδράζονται στην στρατηγική της Ευρώπης 2020 για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και έχουν σαν σκοπό να προωθήσουν την εξυγίανση του τη δημοσιονομική εξυγίανση, να διορθώσουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και να εξασφαλίσουν μια χρηματοοικονομική σταθερότητα. Όλες αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Το σύμφωνο για το ευρώ, το οποίο συμφωνήθηκε από τις επικεφαλείς των κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, ε, και είναι ανοιχτό προς όλες τις χώρες μέλη που επιθυμούν να προσχωρήσουν, αντανακλά ή μάλλον περιγράφει τις δράσεις προτεραιότητες της ε, ετήσιας μελέτης ανάπτυξης. Επίσης αναγνωρίζει το έργο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχέση με την φορολόγηση και την οικονομική ρύθμιση. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω των θέσεων που έχει λάβει και τα πολύ σημαντικές, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις γνωρίσει και να τη συμπεριλάβει. Ε, αυτό ισχύει και για την ε, φορολογική και οικονομική ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή η Οικονομική Επιτροπή επεξεργάζεται μία πρόταση για ε, επιβολή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Και θα ακολουθήσουν δύο συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αποφασίστηκε την περασμένη εβδομάδα, και παρθέτω το απόσπασμα, κρίνοντας ε, τα βήματα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Συμβούλιο αναμένεται να ακολουθήσει τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να εξηγήσει γραπτά τη δική του θέση, τέλος του αποσπάσματος. η να εξηγησει γραπτα τη δικη του θεση τελος του αποσπασματος δημοσιονομική εξυγίανση δεν είναι αυτός σκοπό. Χωρίς δημοσιονομική εξυγίανση δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχουν επενδύσει χωρίς επενδύσεις δεν ε, υπάρχει κανένα ε, είδου ε, ανάπτυξη. Ο στόχος μας όμως, όπως ε, είπα σε αυτό το κοινοβούλιο κατά επανάληψη, είναι η ανάπτυξη, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Και για να το πετύχουμε θα πρέπει να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να ολοκληρώσουμε την ιστορική αγορά. Και ένα από τα προβλήματα που έχουμε εδώ είναι οι διαφορετικές φορολογικές βάσεις. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει και έχει καταθέσει μία κοινή εσωτερική ενοποιημένη φορολογική βάση. Γιατί θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Και η Επιτροπή θα υποβάλει ε, μια, την, μια ενιαία νομοθετική πράξη για την αγορά μαζί με 10 προτάσεις προτεραιότητες προκειμένου να επενδύσουμε στην εργασία και την δημιουργία, ε, προκειμένου να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επίσης, ε, σε στενή συνεργασία με τις χώρες ε, μέλη, η Επιτροπή οριστικοποιεί τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα σύγκλησης σταθερότητας. Αυτό είναι απολύτως ε, σημαντικό για, το, για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εναπόκειται λοιπόν σε κάθε χώρα μέλος να επιτελέσει μια σοβαρή εργασία η οποία να κληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για όλες τις ε, προσπάθειες που οδήγησαν σε ένα πετυχημένο συμβιβασμό όσον αφορά το νομοθετικό πακέτο της Επιτροπής σε σχέση με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει σε μια ε, στεναρή υποστήριξη εκ μέρους της Ευρωβουλής και ελπίζω ότι θα έχουμε μια τελική συμφωνία τον Ιούνιο. Τότε θα μπορέσουμε να εκπονήσουμε ένα νέο οικονομικό πλαίσιο και όλα τα εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς καθώς και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης μέχρι το 2012. Ε, την περασμένη εβδομάδα οι Υπουργοί Οικονομίας συμφώνησαν να δημιουργήσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας από τον Ιούνιο του 2013 με μια πραγματική δανειοδοτική ικανότητα 500 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό βήμα προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία προσπαθεί να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολουθώντα δικέ μα ε, προτάσει, το κείμενο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα ξεκάθαρα τονίζει τον κεντρικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία, καθώ και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την ε, ύπαρξη κινδύνων για την οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης το σύνολό της και να αναλάβει μια ανάλυση της βιωσιμότητας, διατηρησιμότητας του δημοσίου χρέους, το ε, εν λόγω κράτους. Επίσης, αναπόκειται στην Επιτροπή να λάβει ένα ηγετικό ρόλο στην αξιολόγηση των πραγματικών οικονομικών αναγκών του ε, κράτους αυτού, του δικαιούχου κράτους καθώς και την φύση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. Εναπόκειται στην Επιτροπή να προτείνει προς το Συμβούλιο μία απόφαση που να ενισχύει το μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής. Η Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Νομισμό Νομισματικό Ταμείο και μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι υπεύθυνη για την επιτήρηση του βαθμού συμμόρφωσης με, ε, με τους όρους που απαιτούνται, που προϋποθέτουν τα μακροοικονομικά προγράμματα προσαρμογής. Ε, το άρθρο 136 της Συνθήκης διευκρινίζει τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πλαισιωθούν αυτοί οι όροι της οικονομικής πολιτικής, της αποφάσεις του Συμβουλίου και να εξασφαλιστεί μια συνεκτικότητα με το πολυμερές ε, πλαίσιο εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια τακτική βάση σε σχέση με την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ε, νομίζω ότι τελικά πετύχαμε μια συμφωνία η οποία είναι απόλυτα συμβατή με την προσέγγιση της κοινότητας και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την ε, συμμετοχή του σε αυτή την προσέγγιση. Οι χώρες ε, μέλη ε, αναγνωρίζουν την αλεξάρτηση των οικονομιών τους. Αλλά και εδώ θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα ε, ένα υγιές ευρωπαϊκό σύστημα είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. Ένας επόμενος γύρος ε, ε, ελέγχων αντοχής των ευρωπαϊκών τραπεζών θα γίνει τους επόμενους μήνες από την νεοσυσταθήσα Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Η διαφάνεια εδώ είναι απολύτω σημαντική, ούτως ώστε οι επενδυτές να μπορούν να, έχουν, να είναι ενημερωμένοι και να λαμβάνουν, λαμβάνουν τις αναγκαίες αποφάσεις. Ε, ε, ε, θα, θα ήθελα να σας πω ότι παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τον ευρωπαϊκό συντονισμό στην κλιμάκωση της κρίσης στα σύνορα της Λιβύης. Έχουμε ε, κινητοποιήσει 30 εκατομμύρια ευρώ για να παράσχουμε συνδρομή στους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες και έχουμε διάφορες ομάδες επιτόπου και έχουμε στενές επαφές με τις χώρες προέλευσης και τους δωρητές. Ο μηχανισμός ε, προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης συνεχίζει να υποστηρίζει τις χώρες μέλη και τις επιχειρήσεις τους ε, ενώ η δράση σε σχέση με την, ε, με την ζώνη απαγόρευσης ε, πτήσεων εφαρμόζουν το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1973 και θα, και σίγουρα έφεραν ελπίδα στον λαό της Λιβύης και θα μας βοηθήσουν να σώσουμε περισσότερες ανθρώπινες ε, ζωές. Όταν ασχολούμεθα με τους βραχυπρόθεσμους προκλήσεις μιας κατάστασης που αλλάζει ραγδαία, δεν θα πρέπει να χάνουμε από τα μάτια μας το μακροπρόθεσμο στόχο μιας δημοκρατικής, σταθερής και ευημερούσας νότιας Μεσογείου, η οποία να βασίζεται στην ε, εταιρική σχέση που έχουμε προτείνει υπέρ της δημοκρατίας και της ευημερίας. Ο μηχανισμός προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντονίζει επίσης την απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αίτημα της Ιαπωνίας για συνδρομή. Ε, μετά τα γεγονότα της, στην Ιαπωνία προτείναμε να αναθεωρήσουμε την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών και να γίνει μια περιεκτική αξιολόγηση των κινδύνων και να γίνουν έλεγχοι αντοχή σε όλε τι πυρηνικέ εγκαταστάσει στην Ευρώπη. Αυτοί οι έλεγχοι θα πρέπει να διεξαγάγονται επίση σε όλε τι γειτονικέ χώρε και <clears throat> ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικυρώσει αυτό το προσανατολισμό και θα τον ενισχύσει. Εξάτομα μέλη, όπως βλέπετε, έχουμε μια πολύ περιεκτική ημερήσια διάταξη και η Κομισιόν εργάζεται σκληρά προκειμένου να διαμορφώσει σωστά αυτή την ε, ανταπόκριση, αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την οικονομική κατάσταση αλλά και την κρίση στα σύνορά μας. Ε, παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την οικονομική κρίση. Θα το κάνουμε πάντοτε υπό το πνεύμα σεβασμού τη συνθήκη τη Λισαβόνα, που προποθέτει μία συνεργασία με του γείτονέ μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρου των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Πρόεδρος Ζώσεφ Ντόλ που μιλάει εκ μέρους του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ετοιμάζεται να συνεδριάσει για δεύτερη εβδομάδα συνεχεία σε ένα κλίμα βεβαιότητα και διεθνού εντάσεων. Αβεβαιότητα στην Ιαπωνία που ανθρώπινε απώλειε είναι σημαντικέ και εξακολουθούν, είναι δύσκολο να δούμε ακριβώ πόσο είναι. Αβεβαιότητα στη Μεσόγειο όταν εξηγείται νέο λαό κατά του καθεστώτου και στην Ιεμένη και στο Μπαχρέιν. Όλα αυτά έχουν συνέπειε για εμά του Ευρωπαίου. Ε, το δράμα της Ιαπωνίας το ζήσαμε, το ζήσαν άμεσα οι πολίτες μας και υπέφεραν με χιλιάδες οικογένειες που υπέφεραν από το πένθος και επικρατεί ακόμα τώρα που συζητάμε ο φόβος όσον αφορά τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα της Φουκοσίμα και ο φόβος τον ίδιο τον κινδύνο που μπορούμε να διατρέξουμε εμείς σε παρόμοια περίπτωση ή κάτι παρόμοιο ή κάτι το ίδιο θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλε τι χώρε αυτά τα γεγονότα που έχουν πυρηνικού αντιδραστήρε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διοργανώσει συζήτηση όσον αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, χωρί να λιμονούμε την ανάγκη που υπάρχει εμεί οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουμε και όχι να μειώσουμε την ενεργειακή μα ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε από αυτού του θέματο κατά τη διάρκεια τη επόμενη συνόδου μα. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 θα τέλο εβδομάδα συζητήσουν επίση την παρέμβαση αποφάση ΟΗΕ στην Λιβύη για τη διαφύλαξη εκείνων που εξεγέρθηκαν από τι άμεσε ε, επιθέσει του καθεστώτο. Είναι οι ευρωπαϊκέ χώρε, υπογραμμίζω, που ανέλαβαν την πρωτοβουλία αυτών των επιχειρήσεων και που ήταν οι πρώτε να παρέμβουν στην περίπτωση που έπρεπε να υλοποιηθεί η εντολή του ΟΗΕ κατόπιν πρωτοβουλία διαφόρων χωρών ευρωπαϊκών. Και ακούσαμε να το αναφέρουν στην μήνυ σύνοδο, να το αναφέρουν πολλοί συνάδελφοι εδώ στι Βρυξέλλε. Θέλει η ομάδα μου το Συμβούλιο να είναι ευκαιρία για να τελειοποιήσουμε ευρωπαϊκή στρατηγική για τη Μεσόγειο ε, να έχουμε πάντα σαν μέρημνα να βοηθήσουμε και να συνοδεύουμε χωρίς ποτέ να επιβάλλουμε. Είναι δικό μας καθήκον σαν γείτονε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι, μετά σύνοδο κορυφή τη Ευρωζώνη περασμένη εβδομάδα που ετοίμασε το έδαφο και τα μέτρα φάρου για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι τρει εβδομάδε αυτά τα μέτρα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του ευρώ και τη βελτίωση τη οικονομική διακυβέρνηση. Η ομάδα του ΕΛΚ είναι υπέρ τη αύξηση των πόρων που διατίθεται για την υποστήριξη του ευρώ και για τη διόνυση των μέσων ad hoc που ε, θεσπίσαμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Αυτή η πολιτική βούληση ε, δείχνει πόσο επέφθυνα τα κράτη-μέλη στον αφορά τη διαχείριση μια κρίσης άνευ προηγουμένου από τη δημιουργία του ενίου νομίσματός μας. Επιμένουμε στεναρά όμως ε, ώστε η εξαιρετική αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε από την παρέκκληση των εθνικών δημοσιονομικών να μην είναι μια ευκαιρία για το Συμβούλιο να αλλάξει μέθοδο όσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Η κοινοτική μέθοδο θα πρέπει να παραμένει ο κανόνος και η διακυβερνητική μέθοδο η εξαίρεση. Υπάρχει μια πλειοψηφία πολύ μεγάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποστηρίζει αυτή την αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μπαρόσο υποστηρίζει σε αυτό το διάβημα διότι είναι ζωτική σημασία για την εξέλιξη τη Ένωση και το μέλλον. Δεν αμφισβητώ ότι ο πρόεδρο Βαν Ρομπόη θα μπορέσει να πει στου αρχηγού και κυβερνήσεων για αυτό το θέμα. Την Παρασκευή θα πρέπει επίση να υιοθετηθεί και το σύμφωνο για το ευρώ. Ένα σύμφωνο που υποδεχόμαστε θετικά στο βαθμό που προβλέπει αυτό που ζητούμε εδώ και μήνε. Δηλαδή, ε, μια σύγκληση των δημοσιονομικών πολιτικών, των κοινωνικών και των φορολογικών μεταξύ κρατών μελών. Το λέω και το επαναλαμβάνω. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν θα γίνει αποδεκτή από του λαού μα παρά μόνο αν το θεωρεί ότι είναι κάτι που το αξίζουν και δίκιο. Αυτό δεν θα ισχύσει παρά μόνο αν συνθήκε εργασία πληρούνται και αν οι επιχειρήσει μα μπορούν να επενδύουν και να προσλαμβάνουν σε ένα περιβάλλον φορολογικό συγκρίσιμο. Τέλο, η ομάδα μα ζητά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσει γρήγορα, το Συμβούλιο να προχωρήσει γρήγορα όσον αφορά το πακέτο τη οικονομική διακυβέρνηση και να λάβει δόντω υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι συνομοθέτη σε τέσσερα από τα έξι χαρτοφυλάκια που συζητούνται. Η Ευρώπη θα πρέπει να ξαναβρει το μονοπάτι τη ανάπτυξη και τη απασχόληση και τα μέτρα που σχεδιάζονται πάνε προ σωστή κατεύθυνση. Όμω, εν τούτης, ό,τι και αν αποφασιστεί σε ένα κοινοτικό πλαίσιο, ε, θα πρέπει να επιτρέψει στην Ευρώπη να ε, συνεχίσει τη συζήτηση για αυτά τα θέματα και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο κύριος Πρόεδρος Μάρτιν Σούλτς έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θερμά συγχαρητήρια για τα σημερινά σας γενέθλια. Χρόνια σας πολλά. Έχετε κάθε απέτηση να τύχετε συγχαρητηρίων για τα γενέθλιά σας. <laughs> Επιμένω και εμένα τα 15 δευτερόλεπτα για τα χρόνια πολλά να αφαιρεθούν από το χρόνο που έχω ως ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται υπερβολική ευγένεια έναντι του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορώ να, συ, να συμμεριστώ την δική σας ικανοποίηση ενώπιον αυτής της Συνόδου. Νομίζω ότι είναι στη χειρότερη φάση, υπό τους χειρότερους όρους και προϋποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αυτή η Σύνοδος Κορυφής. Ξεκινά με τη Λιβύη. Σπάνια είναι μια δράση τόσο βιαστική και τόσο χωρίς σωστή διάρθρωση όπως αυτή στην Λιβύη που υποτίθεται ότι θέλει να βοηθήσει ανθρώπους αλλά που σε σχέση με την έκβασή της ελπίζω να μην έχει ολέθρια έκβαση χωρίς συντονισμό και χωρίς συντεταγμένη διάρθρωση η Ευρώπη κινείται προς ε, κάθε κατεύθυνση και η υποψήφια ένταξη Τουρκία τροχοπερεί τα πάντα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν όπου πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε αυτή την κρίση. Εδώ και ένα χρόνο η ίδια διαδικασία λειτουργεί και συνεχίζεται. Αυτά τα οποία είναι αναγκαία καταρχήν ε, δεν υλοποιούνται ώστε με ολόκληρη μεγάλη καθυστέρηση να κάνουμε κάτι. Οι Έλληνες να αυτοβοηθηθούν λέει ε, και μετά από τέσσερις μήνες τι έγινε μηχανισμός διάσωσης της Ελλάδα. Δεν χρειάζεται κάποια ομπρέλα διάσωσης ε, λέγεται. Μετά από τέσσερις μήνες τι βλέπουμε χρειάζονται περισσότερα χρήματα παρόλα αυτά. Δεν θέλουμε ευρωομόλογα. Είναι ανοησία λέει τα ευρωομόλογα. Η συζήτηση για τα ευρωμόλογα προ κάθε κατεύθυνση διεξάγεται. Και θα έρθουν, θα υιοθετηθούν τα ευρωμόλογα σίγουρα, αλλά με καθυστέρηση τεσσάρων μηνών. Δεν χρειάζεται οικονομική διακυβέρνηση, λέει. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη οικονομική διακυβέρνηση. Οι ίδιοι άνθρωποι που τα λένε αυτά και που ισχυρίζονται αυτά ε, με κάθε τρόπο τώρα χαιρετίζουν την ε, διακυβέρνηση που θα υιοθετηθεί και δεν τρέπονται που κάνουν το αντίθετο από αυτό το οποίο τώρα προαναγγέλλεται. Και δεν ξέρω αν η κοινοτική μέθοδος έχει διασωθεί. Το ελπίζω να έχει διασωθεί. Και έχετε την υποστήριξή μας σε αυτό το εγχείρημα κύριε Μπαρόζο. Ναι, όχι ως δώρο γενεθλίων, αλλά επειδή πρέπει να υπερασπιστούμε το κοινό νόμισμα και την νομισματική ένωση και να δούμε με την ενωσιακή μέθοδο να προχωρήσουμε και όχι με άλλες μεθόδους που η κυρία Καγκελάριο Μέρκελ χαρακτηρίζει ω τη νέα ευρωπαϊκή μέθοδο. ακριβώ δηλαδή αυτά τα οποία περιέγραψα πιο πριν. Καθένα κάνει ότι του κατεβαίνει και την επομένη κάνει το αντίθετο αυτόν που είχε προαναγγείλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχουμε κρίση ευρώ μπροστά μα. Έχουμε όμω μια κρίση κυβερνήσεων κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης ευρώ. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Στην Πορτογαλία όλοι συζητούν και μιλούν και ελπίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση που πραγματικά πάρα πολύ σκληρά, πίστευτα σκληρά μέτρα υιοθετεί όπως μια κυβέρνηση όπως και στην Ελλάδα υιοθετεί τέτοια μέτρα εν μέρει και κατά της έγκρισης των ε, πολιτών και βλέπουμε πώς αφήνουμε αυτή την κυβέρνηση να ε, είναι απομονωμένη και μόνη της. Στην ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία ο Υπουργός Οικονομικών που είναι λέει φιλοευρωπαίος λίγες μέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής κλείνει ένα πακέτο μέτρων που το χρειαζόμαστε όλοι και πάει ο Υπουργός Εξωτερικών και η Ομοσπονδιακή Καγκελάρια και λέει όχι αυτό το πακέτο δεν μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει πρώτα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη Παρασκευή να συζητήσω με πάρα πολλού εκπροσώπου του οικονομικού κόσμου στην Ευρώπη για το θέμα αν την χάνει ή όχι το ευρώ τη εμπιστοσύνη. Η απάντηση των υπεύθυνων στην Φραγκφούρτη που συζήτησα μαζί του και μεταξύ αυτών ο πρόεδρο ε, τη ε, Ευρωζώνη, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και πολλοί άλλοι επικεφαλεί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είπαν ναι, το ευρώ είναι ένα σταθερό νόμισμα την χάνει εμπιστοσύνη στο ευρώ και έχουμε και εμείς εμπιστοσύνη στο ευρώ. Όμως δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που στηρίζουν αυτό το ευρώ. Διότι πώς θέλει κανείς να έχει εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που δεν κρατάει τον λόγο της ούτε για τρεις μέρες όλες και όλες. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη σήμερα και πρέπει να καταπολεμήσουμε. Η πορεία είναι λανθασμένη. Το ευρώ είναι ένα ισχυρό νόμισμα το ευρώ είναι η έκφραση της ε, ρόμης και δύναμης της Ευρώπης εναντί των άλλων υπήρων το ευρώ από την εισαγωγή του είχε ένα δολάριο 17. Τώρα κοιτάξτε πόσο έχει το ευρώ. Είναι ένα σταθερό νόμισμα διπυρωτικά στον ανταγωνισμό των νομισματικών ζωνών το ευρώ. Αλλά εσωτερικά αποσταθεροποιείται επειδή δεν υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις με σταθερή πορεία. Γι' αυτό η κοινοτική μέθοδος δεν είναι μόνο αντικείμενο συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τα θεμέλια για τη σταθεροποίηση του νομίσματος του νομίσματος που είναι έκφραση τεράστιας δύναμης και δυναμικού της Ευρωζώνης. Μόνο που αυτό το δυναμικό, αυτή η δύναμη οικονομική δεν μπορεί να απελευθερωθεί επειδή την διοικούν και την διακυβερνούν ε, πολιτική που για αυτούς έχει μεγαλύτερη σημασία η εκλογική αναμέτρηση σε κάποια περιφέρεια της χώρας τους ε, και όχι το στο ευρώ. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω τα όσα προαναγγείλατε να επισυμβούν, να ε, γίνουν πραγματικότητα. Ελπίζω με θετικά μαντάτα έχουμε την ολοκλήρωση της Συνόδου. Όμως ειλικρινά φοβούμε ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε αυτό που ζούμε εδώ και ένα χρόνο κιόλα. Λυπούμε, πρέπει να το πω έτσι ξεκάθαρα. Πραγματικά δηλαδή, εδώ <clears throat> είναι πρόβλημα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος θα έχει τώρα για 4,5 λεπτά. Euh, συγχαρητήρια στον πρόεδρο Μπαρόζο όπως και εγώ η Μαρία Σαρνές και ο Τζόσεφ Ντόιλ, εδώ έχουμε πολύ... να κρύοι, είμαστε κρύοι. Αλλά έχουμε κάποια σχόλια να κάνουμε όσον αφορά το σύμφωνο αυτό, διότι καλό που όλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη και χρειάζεται οικονομική κυβέρνηση, έχει κεφαλαίου σημασία στο ερώτημα. Το σύμφωνο για, την, για το ευρώ πραγματικά θα δημιουργήσει ένα λέοντα οικονομικό. Αυτό το σύμφωνο θα δημιουργήσει την οικονομική διακυβέρνηση και την Ένωση την οικονομική. Δεν το πιστεύω και για τον απλούστατο λόγο, διότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι επικεφαλή τη ε, διαδικασία. Παραμένουν τα κάτι μέλη παρόλα αυτά και δεν είμαι εγώ αυτό που το λέω, έχω τα κείμενα τη 11 η Μαρτίου. Το κείμενο μάλλον που θα υιοθετηθεί αύριο και μεθαύριο, τα κείμενα μάλλον. Λέει ότι οι στόχοι αποφασίζονται από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Ότι οι δεσμεύσει αναλαμβάνονται από του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων ότι παρακολούθηση γίνεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς κάνει την τεχνική δουλειά, τίποτα άλλο, την τεχνική παρακολούθηση. Όλη η εξουσία είναι στο Συμβούλιο. Και αυτό ήταν ε, το πρόβλημα της στρατηγικής της και το ελάττωμα. Και αυτό θα είναι και η ήττα, θα αποτελέσει την ήττα και αυτή της στρατηγικής. Αυτό που νίξε την στρατηγική της Αβώνας. Γι' αυτό ζητάει άλλη καμιά φορά ε, να προετοιμάσουμε μαζί με τον κύριο το ταχύτερο δυνατό αυτό πρέπει να εγκριθεί. Ένα πραγματικό σχέδιο οικονομική διακυβερνήσεω που θα βάζεται σε κοινοτική πράξη που θα δίνει όλη την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα εδράζεται επί κώδικα σύγκληση και θέτει επιτάπητο του Συμβουλίου τα θέματα. Λένε πάντα όχι, όχι. Συνεχίστε τη μάχη μαζί μας και μη δεχόσαστε αυτή τη διαδικασία και την πρόταση που είναι επιτραπέζη σε αυτή τη φάση, διότι δεν θα λειτουργήσει και θα σταθεροποιήσει το ευρώ του επόμενου μήνε και τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω. Το δεύτερο σχόλιο που έχω, κυρία Πρόεδρε, αφορά την ε, επανάσταση των Αράβων και τη συνέχιση της συζητήσεω που είχαμε εδώ και μια εβδομάδα πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι μπορούμε να κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό της ευρωπαϊκής δράσεως. Και αυτός ο πρώτος απολογισμός είναι θα έλεγα τι να μέτριος. Στην αρχή θα θυμόσαστε πολύ καλά ε, δεν είμαστε πολύ ενθουσιώδεις όταν μιλούσαμε για την επανάσταση των Αράβων. Λέμανε, α, είναι φονταμεταλισμός Ισλαμικός ο οποίος θα καταφτάσει. Το πρώτο πράγμα που κάναμε στις ευρωπαϊκές αρχές, στους ευρωπαϊκούς φορείς, στην ε, Λιβύη, στην υπόθεση Λιβύη, δείξαμε την έλλειψη ένωση Ευρωπαϊκή Ενώσεω και το θεωρώ αυτό φρικαλαιώδες στο Συμβούλιο Ασφαλείας όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω δεν είχαν την ίδια θέση. Υπήρχαν τρεις που ψήφισαν ναι και ένας που απήχε. Και λέω ότι αυτό είναι αντίθετο προς συνθήκε. Στη συνθήκη υπάρχει το άρθρο 34 της συνθήκης που αναφέρει ότι αν σε κάποιο φορέα μιλούμε για την εξωτερική πολιτική, τα κράτη-μέλη της Ένωσης υπέχουν υποχρέωση να συντονίζονται και να έχουν την ίδια άποψη σε αυτό τον φορέα το συγκεκριμένο. Το κάναμε? Δεν νομίζω ότι το κάναμε και ότι παραβιάσαμε μάλιστα και το άρθρο 34 της συνθήκης. Και μετά, τρίτον, αυτό που βλέπω τώρα και λυπούμε που το λέω. Χθε η κυρία Άστον ήταν στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα επίση, όταν μιλάμε για ένα θέμα τόσο σημαντικό. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει έλλειψη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι επαναστάσεων στι αραβικέ χώρε. Αυτό που βλέπουμε να απορρέει από τι αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καμιά φορά σκανδαλώδε. Την Παρασκευή, παραδείγματο χάρη, στην ΑΦΕΤ ήταν τη Δευτέρα ο κύριο Κούπολ που είναι ένας από τους συνεργάτες της κυρίας Άστον είπε σε κάποια δεδομένη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε την κατάσταση στο Μπαχρέιν και οι αρχές είχαν δίκιο να θέλουν να αποκαταστήσουν την τάξη και την ηρεμία. Τη στιγμή που είχαν σκοτωθεί τέσσερα άτομα και 200 τραυματιστεί. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή θέση. Είπα το χάρη για να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Υπουργό Εξωτερικών της Ενώσεως οι Υπουργοί Εξωτερικών Συνεδριάσεω συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τι είπαν, εκάλεσαν επίση, και μιλάω για τον Μπαχρέιν, του διαδηλωτέ να απόσχουν από κάθε πράξη ε, σκόπιμη ε, πίεσης και πρόκλησης αντί να υποστηρίξουμε αυτή την επανάσταση και εκείνους που είναι στους δρόμους, αυτούς που πολέμησαν, αυτούς που σκοτώθηκαν, γιατί αυτό που κάνουν, το αντίθετο κάναμε. Λέμε μείνετε ήρεμοι, προσέξτε, αυτό που ζητώ είναι η κυρία Άστον να έρθει στην Ολομέλη. Αυτό ζητώ. Να εξηγήσει ποια είναι η στάση, ποια είναι η στρατηγική που θέλει να ακολουθήσουμε. Στον Παχρέιν, στη Συρία, στην Ιεμένη. Ποιε είναι οι κυρώσει που θέλουμε να εφαρμόσουμε και με ποιον θα το κάνουμε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε παρά να κάνουμε αυτές τις αξιοθρύνητες τοποθετήσεις πολλών από τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Σαχραντήλ έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπούμε που λέω που βλέπω ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιφέρει κάποιου πραγματικούς κινδύνους και θα πρέπει να ανησυχήσουμε γι' αυτό. σε σχέση με τον οικονομικό συντονισμό, την οικονομική διακυβέρνηση, τη σταθερότητα για την Ευρωζώνη, βλέπουμε εύνοια όσον αφορά την, τον εναρμονισμό των φόρων και ένα ενιαίο πλαίσιο και το Κοινοβούλιο έχει δυστυχώς ε, διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο για όλα αυτά. Ας το πω ξεκάθαρα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για μια κοινή παγία ε, θέση όσον αφορά την φορολόγηση θα είναι επιζήμια για την οικονομία, για τον ανταγωνισμό και θα διώξει τις επιχειρήσεις από την Ευρώπη σε σχέση με αυτούς που θα επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Όλα αυτά πάνε πολύ μακριά και πρέπει να σταματήσουν. Αυτά τα οποία είδαμε τις τελευταίες ήταν μια προσπάθεια απόπειρα από τα κράτη-μέλη να αναμειχθούν στα θέματα φορολογίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων των άλλων κρατών μελών. Γνωρίζετε γιατί πράγμα κάνω λόγο για κάτι πραγματικά ατυχές ε, το θέμα αυτό επιβολή στην Ιρλανδία αυτών των ε, κελευσμάτων πιθαναγκαστικά. Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί. Οι εξελίξεις στη Λιβύη μας υπενθύμησαν για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να αναμένουμε υπερβολικά πολλά από την αποκαλούμενη κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας. Οι εθνικοί ηγέτες ε, έχουν δείξει ηγετικό πνεύμα. Ο Πρωθυπουργό Κάμερον και ο Πρόεδρος Σαρκοζή επέβαλαν αποφάσεις και όχι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δείχνει με σαφήνεια ότι υπάρχουν όρια όσον αφορά την ολοκλήρωση σε αυτό το επίπεδο και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο. Κανένα κράτος μέλος δεν θα έπρεπε να αισθάνεται υποχρεωμένο να κάνει περισσότερα από αυτά που θεωρεί αναγκαία. Και πρέπει αυτό να το δούμε σε σχέση με την εξωτερική πολιτική αλλά και την οικονομία. Πρέπει να είναι ευέλικτη η Ευρώπη όπου είναι δυνατόν και να μην έχουμε άκαμπτα δόγματα ολοκλήρωσης. Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή της πολιτικής ε, του υποδείγματος που ακολουθείται για την ολοκλήρωση. Είναι σαφές κατανοητό αυτό και ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα το λάβει υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτς έχει το λόγο τώρα για την ομάδα των Πρασίνων για δυόμιση λεπτά. Ε, πρόεδρε, ο κύριος Μπαρόζο δεν βρίσκεται πλέον εδώ, αλλά είπε ότι η εμπιστοσύνη είναι η βάση των πάντων. Θα ήθελα να σας πω ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών μας εξατμίζεται τόσο γρήγορα όσο το νερό στη Φουκουσίμα. Ναι, υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πλέον όπως το παρελθόν. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα και λιγότερη επισφάλεια. Θα πρέπει να ε, εμπιστευτούμε την οικονομία και η οικονομία θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη. Δεν είναι δυνατόν να οικοδομούμε πλέον την οικονομία μα ε, στο χρέο, είτε πρόκειται για ιδιωτικό είτε για δημόσιο χρέο, είτε στα ελλείμματα και στην κερδοσκοπία. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι πολίτε μα και οι συμπολίτε μα γνωρίζουν ότι όλα αυτά συνεπάγονται ριζοσπαστικέ αλλαγέ εκ μέρου των κυβερνήσεων, εκ μέρου των επιχειρήσεων και εκ μέρου των ιδίων. Το γνωρίζουν και το διαισθάνονται και διαισθάνονται ότι αυτέ οι ριζοσπαστικέ αλλαγέ είναι σύνθετε και συνεπώ δεν μπορούν να γίνουν όλα δια μια. Θα πρέπει κάπου να ξεκινήσουμε. Αλλά βλέπετε για του συμπολίτε μα ε, πάντοτε αρχίζουμε από το ίδιο σημείο. Ε, πάντοτε από την περικοπή των δημοσίων δαπανών. Ε, και αυτό γίνεται σε βάρος των πιο αδυνάμων. Η αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο ευέλικτη. Από εκεί ξεκινάμε. Γιατί όταν μιλάμε για την Security ε, πρόκειται για περισσότερη ευελιξία και λιγότερη ασφάλεια. Τώρα, αυτό το οποίο αναμένουμε από το Συμβούλιο είναι από τη μία μια τολμηρή πρωτοβουλία που να εξασφαλίσει τις χώρες μέλη ε, δημοσιονομικά έσοδα και σταθερά έσοδα μέσω της φορολόγησης των χρηματοπιστικών συναλλαγών, της ενέργειας και επιβολής ε, φόρου στις επιχειρήσεις. Ε, δεν είναι δεδόν πλέον να συνεχίσουμε με αυτό το φορολογικό νιρβάνα. Επίσης, πάλι κατά των φορολογικών παραδείσων. Μπορώ να σα πω ότι όλα τα θέματα που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση ε, θα καταρρεύσουν γιατί δεν υπάρχει ιστορικό παράδειγμα μιας νομισματικής ένωσης που να έχει πετύχει χωρίς ε, μια δημοσιονομική ε, στεναρή ένωση. Τώρα, δεν είναι τα νέα stress test τα οποία θα μας φέρουν περισσότερη ασφάλεια ούτε στους πυρηνικούς σταθμούς. είδαμε τι έγινε με τα προηγούμενα stress αυτό που χρειάζεται είναι νέοι δεσμευτικοί κανόνες. Όχι οι κανόνες που λέμε ότι θα ελοπιθούν το 2019. Είναι σημαντικό σήμερα ε, να τεθούν κάποια όρια, γιατί οι συμπολίτες δεν μπορούν πλέον να περιμένουν. Και μόνο με τον τρόπο αυτό θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που είναι αναγκαία για να μας επιτρέψει εμάς τους Ευρωπαίους να έχουμε το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία του τον 21ο αιώνα ο κύριος της ε, Ευρωπαϊκή Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια οικονομική και νομισματική ένωση χωρίς ε, αποτελεσματικό οικονομικό συντονισμό δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει αποτύχει και ε, σε αυτό το σημείο πολλοί ειδικοί πέρα από τα, πολιτικά, τα όρια των πολιτικών ομάδων συμφωνούν. Πράγματι δεν είναι ορατά στον ορίζοντα νέα πολιτικά μοντέλα. Το 3% όριο του Συμφώνου Σταθερότητας έχει θεσπιστεί, δεν έχει τηρηθεί από το 1999 και 46 φορές δεν θα ήταν ανεκτό και καμία φορά δεν έχει επιβληθεί κάποια κύρωση. Τώρα δεν θα αλλάξει το μη εφαρμοσμένο σύμφωνο σταθερότητας, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί καλύτερα. Όλοι βεβαίως γνωρίζουν, όλοι οι επιχειρηματίες γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι ένα ε, βιώσιμο προπολογισμό. Όσον αφορά τι αποφάσει για την οικονομική διακυβέρνηση και για τον, οικονομικό, για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα, ε, φοβούμεθα ότι εδώ ο σκοπό είναι μόνο η εξοικονόμηση ε, πού βρίσκεται η βιωσιμότητα. Καμία χώρα η οποία είναι τόσο χρεωμένη, που βρισκεται η δυοσημοτητα καμια χωρα η οποια ειναι τοσο χρεωμενη που βρισκεται στα όρια της ε, χρεοκοπίας, δεν είναι το να εξαλειφθεί την παγίδα του χρέους εάν ε, συνεχίσει να δανείζεται ε, με πολύ ψηλά επιτόκια. Όσο και αν εξοικονομεί, το χρέος διονγκούται και διονγκούται πολύ περισσότερο εάν οι συντάξεις και οι μισθοί συρρυκνώνονται αλλά οι επενδύσεις και επενδύσεις στην παιδεία, στην υγεία κλπ. επίσης ε, υποχωρούν, συρρυκνούνται. Ε, εκεί που δεν υπάρχει ζήτηση και κατανάλωση μειώνεται η οικονομία. Ούτε η όξυνση του συμφώνου σταθερότητας, ούτε η επιβολή κάποιων αυστηρών όρων στο πλαίσιο του μηχανισμού σταθερότητας θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα και τα δύο είναι παραπλανητικά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε πιο ξεκάθαρα είναι επισήμανση μιας ανάγκης επιπλέον επενδύσεων, ιδιαίτερα σε χώρες που απειλούνται από την κρίση και μάλιστα μέσω, με την, μέσω επιμήκυνσης των, της διάρκειας των δανείων και μίας των επιτοκίων. Αλλιώς η κατάσταση θα είναι προβληματική γιατί απαιτούνται ε, λήψη μέτρων μόνο από τις οικονομικά δύναμες χώρες, ενώ οι πλούσιες χώρες συνεχίζουν όπως και στο παρελθόν. Και τα ε, ελλείμματα ε, των μεν τελικά δεν είναι τίποτα άλλο, των αδημάτων δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλεονάσματα των δυνατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα όσα μας ανήκει λέει ο κύριος Μπαρόζο αποτελούν μια ουσιαστική πρόταση για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και της σταθερότητας του ευρώ. Αυτό σημαίνει η επιτάχυνση της πολιτικής και οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Βέβαια, η εργασία του κυρίου Μπαρόζο, που συνεπικουρείται από τον κύριο Όλι είναι πάρα πολύ επιτυχής και την βλέπουμε θετικά ελπίζουμε δε να μπορέσει να ανταποκριθεί το σύμφωνο αυτό στις οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις της ένωσης και να στείλει το μήνυμα που πρέπει τις αγορές. το πρόβλημά μας δυστυχώς σήμερα έχουν γίνει οι αγορές. η νέα οικονομική διακυβέρνηση έρχεται μετά από μια κρίση μια βάναυση κρίση του δημοσίου χρέους των κρατών μελών. βεβαίως κατά την άποψή μου όταν οι ηνωμένε πολιτείε εκδίδουν νέο νόμισμα που υπολογίζεται σε πάνω από 3, εκατομμύρια δολάρια δεν βλέπω γιατί η ευρώπη δεν μπορεί να δώσει τη λύση με έκδοση ενός ε, νέου νομίσματος της τάξης του 1 τρει ευρώ το οποίο να μην μπει στην αγορά αλλά να αποτελέσει κεφάλαιο αυτό που λέμε ε, μηχανισμό στήριξης. Εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι δεν είναι όριμες αυτές οι σκέψεις να περάσουν υπό το καθεστώς της κυρίας Μέρκελ κυριαρχούσης στην Ευρώπη όμως για άλλη μια φορά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ευρωπαϊκή ένωση αναγκάζεται να προβεί στη δημιουργία νέων συστημάτων και αξιών κάτω από αντίξωες συνθήκες και υπό αναγκαστική κατάσταση. η ύπαρξη νομισματικής ένωσης χωρίς τη συνολική στρατηγική οικονομικής διακυβέρνησης και συντονισμού των κρατών μελών ήταν ένα ρίσκο που δοκιμάστηκε στην πράξη και λειτουργήσε σε γενικές γραμμές ήρθε η ώρα η ένωση να πάρει πιο γενναίες αποφάσεις πιστεύω και να κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει. οι αποφάσεις του συμβουλίου βεβαίως για το σύμφωνο του ευρώ μας βρίσκουν όπως είπα κατά βάση σύμφωνους και θεωρούμε ότι το ευρώ θα συνεχίσει να αποτελεί ένα καλό νόμισμα. όμως κυρία πρόεδρε θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο στόχος όχι μόνο η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ αλλά και η εξασφάλιση υψηλού επίπεδου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην ευρώπη η αύξηση και διατήρηση των θέσεων εργασίας των ευρωπαίων πολιτών και κυρίως των νέων. πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στους νέους. ευχαριστώ. ο κύριος Μάρτιν εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ως διακαής ευρωπαϊστής και θα έλεγα και σαν τη μεγάλη πλειοψηφία των 500 εκατομμυρίων πολιτών είναι πολύ δύσκολο αυτή την δύσκολη κατάσταση στην οποία καταλήξαμε να την δεχτούμε. Από τη μία πλευρά λέμε ναι σίγουρα, μάλιστα χρειαζόμαστε τη σταθερότητα. Κάτι πρέπει να κάνουμε κατά της κερδοσκοπίας. Από την άλλη πλευρά ο τρόπος όπως προωθούνται αυτά και πάλι είναι μια αφορμή το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δραστικό τρόπο να καταδεικνύεται και πάλι. Ο τρόπος υπενθυμίζει περισσότερο διατάγματα έκτακτης ανάγκης ε, και όχι αυτά που επιθυμεί κανεί από μια ανεπτυγμένη Ευρώπη. Γι' αυτό έχουμε υποστηρίξει την τροπολογία 34 της ενωτική Αριστεράς των Αριστερών που απαιτεί, ζητεί την υιοθέτηση της κανονικής αλλαγής της συνθήκης. Και πού καταλήγουμε, σε μια κατάσταση ανάγκης όπου το χάσμα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται διαρκώς. Και κατά τα άλλα θα ήθελα να πω ότι αυτά τα οποία είπε ο Μάρτιν Σούλτσα τα απορρίπτω και μάλιστα κατηγορηματικά. Ευχαριστώ. Τελείωσαν οι παρεμβάσει εκ μέρου των πολιτικών ομάδων και ερχόμαστε στου άλλου εγγεγραμμένου ομιλητέ. Ο κύριο Σαλαφράγκα για δύο λεπτά, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κρίση στη Βόρεια Αφρική αποτελεί δοκιμασία για τους μηχανισμούς της συνθήκης Λισαβόνας. Χθες, στην παρουσίαση της της εκπροσώπου στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, υπογραμμίσαμε τις θετικές πτυχές της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανακοίνωση της κυρίας ε, Άστον που διαφοροποίησε μεταξύ βραχυπρόθεσμων και ε, μακροπρόθεσμων μέτρων, ε, ταχεία υιοθέτηση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο και δράση δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σωστό να τίθενται όλα αυτά, αλλά όμως υπάρχουν ερωτηματικά από πλευρά των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό οι πολίτες μας, κυρία προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Ο κύριος Φερχόφστατ για αυτούς τους λόγους έχει απόλυτο δίκιο. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χρονική στιγμή τα τέσσερα κράτη-μέλη που αποτελούν με, τμήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να μην ψηφίζουν με τον ίδιο τρόπο, να ψηφίζουν διαφορετικά. Πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χρονική στιγμή να συζητάμε αν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών θα το εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το εφαρμόσει το ΝΑΤΟ ή η Διεθνή Συμμαχία, όταν κάνουμε λόγο για τους ίδιους πόρους, που προέρχονται από του ίδιου ε, εισφορείς, ε, από του ίδιου φορολογούμενους ε, και χρησιμοποιούνται τα ίδια πλοία στο ίδιο θέρετρο επιχειρήσεων. Πολλά έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την ικανότητα συντονισμού μας και πολλά πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Υπάρχει μια γνωστή φράση από ένα έργο, την Καζαμπλάνκα, που λέει πάντα θα έχουμε το Παρίσι. Και γι' αυτό η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μια πολύ βιαστική απάντηση πρέπει να πούμε. Αν δεν ήταν το θάρρος, η στεναρότητα και η συνεκτικότητα και ε, συνοχή της Γαλλίας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό ξεκάθαρα αναγνωρίζοντας ε, τους επαναστάτες της Λιβύης ε, αποστέλλοντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το θέμα και εφαρμόζοντας το ψήφισμα <clears throat> των Ηνωμένων, του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών, οι στρατιωτικέ δυνάμει του Γκαντάφη θα είχαν εισέλθει ήδη στη Βενγάζη. Ευχαριστώ. Ο είναι, έχει το λόγο για δύο λεπτά, παρακαλώ. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да се концентрирам малко повече върху една. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να εστιαστώ περισσότερο επί ενός από τα καυτά ζητήματα προς συζήτηση αύριο ή κατάσταση στην Ιβή. Πολύ σωστά το ανέφεραν οι προλαλήσαντες ότι οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν σχεδόν χαοτική στάση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από πλευράς των διαφόρων κρατών μελών. Το ότι κάποια κράτη-μέλη πηγαίνουν με τη συμμαχία και μετά θέλουν να αποσυρθούν το γεγονός ότι δεν υπάρχει εμφανή συμφωνία εντός του ΝΑΤΟ, όλα αυτά μαζί με τη σύγχυση που δημιουργούν μεταξύ των εταίρων μας σχετικά με το τι εννοούμε και τι θέλουμε να πετύχουμε, δημιουργεί επίσης μια βεβαιότητα εντός ε, της ευρωπαϊκής κοινή ε, γνώμης και χάνουμε τελικά αξιοπιστία. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα προσδοκόμενα, στα αναμενόμενα στη Νότια Μεσόγειο. Και θα ήθελα να δω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, να προβεί σε μια σαφή, ξεκάθαρη απόφαση τι επόμενες μέρες όσον αφορά τη Λιβύη. Αλλά όχι μόνο τη Λιβύη, Μπαχρέιν μετά, η Εμένη, Συρία σε κάποιο βαθμό. Όπου εκεί έχουμε παρόμοιες εξελίξεις. Κατά κάποιο τρόπο λησμονούμε ότι αυτό που κάνουμε στη Λιβύη θα αξιολογηθεί ε, και εν συγκρίση με το τι κάνουμε σε άλλα μέρη της περιοχής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει πραγματικά να διαπιστώσει τι θέλει να πετύχει στη Λιβύη. Και μόνο άμα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα θα γνωρίσει το Συμβούλιο πώς να πετύχει το στόχο. Και μετά πρέπει να είναι και κάτι άλλο ξεκάθαρο, ότι η κατάσταση στη Λιβύη θα έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις γειτονικές χώρες. Εάν η κατάσταση εξακολουθήσει να ισχύει επί μακρόν στη Λιβύη ως έχει τώρα, πρέπει να βοηθήσουμε επίσης και την Τινησία και την Αίγυπτο, όχι μόνο να ασχοληθούν με την άμεση ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με την ανάκαμψη, την οικονομική ανάκαμψη και μετά αυτή τη φάση. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελέγχθη ότι ε, δεν διακυβεύεται το ευρώ στην κρίση, αλλά οι χώρες ε, μέλη που έχουν κάνει ανεύθυνα, έχουν σφαιρέσει ανεύθυνα χρέη ε, εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει. Είναι ορθό ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας προποθέτει μια αύξηση των ε, πόρων. Είναι ε, ορθό το ότι η Ιρλανδία δεν ε, κέρδισε μια μείωση των επιτεκείων. Ακούω από τους σοσιαλδημοκράτες να γίνεται μια διάκριση μεταξύ καλού και κακού χρέους. Βεβαίως η επένδυση είναι κάτι άλλο από την κατανάλωση, αλλά κάποτε τα υπερβολικά, τα πάρα πολλά καλά χρέη θα μεταβληθούν σε κακά χρέη. Χρειαζόμαστε μια βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας το σύμφωνο για, την, για το ευρώ ε, χωλαίνει όσον αφορά το, ε, την κοινωτική πολιτική. Ε, όσον αφορά τη Λιβύη, ε, συμφωνώ με τον κύριο Σαλαφράκα που είπε ότι ήταν θετικό ο ρόλο τη Γαλλία, αλλά θα έπρεπε να έχει εκλειθεί και η Τουρκία. Και στην περίπτωση αυτή η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο εύκολη στο ΝΑΤΟ. Και ελπίζω ότι ο νέο ε, επικεφαλή τη μεταβατική λιβική κυβέρνηση θα γίνει σύντομα αποδεκτό, θα προσκληθεί σύντομα στην Ευρώπη. Λόγω για ένα λεπτό. ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, όλοι οι στόχοι των χωρών μελών της ζώνης ευρώ, κάποιοι από τους οποίους είναι πολύ καλοί, μπορούν να επιτευθούν μέσω συντονισμού της οικονομικής πολιτικής. Τίθεται όμως ένα ερώτημα εδώ και αυτό είναι γιατί αυτές οι εξουσίες μεταφέρονται, μετατίθενται τώρα σε ενωσιακό επίπεδο θα μπορούσε να είναι ένα θέμα διασποράς ευθυνών όσον αφορά μη δημοφιλής στο επίπεδο των Βρυξελών. Αμφιβάλλω αν αυτά όλα θα επιτύχουν τον ευκταίο στόχο. Η Ευρωζώνη, τα κράτη-μέλη έχουν πάρα πολύ υψηλό χρέος και μη ανταγωνιστικές οικονομίες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Δημιουργείται εδώ λοιπόν μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, με άλλα λόγια. Η ταχύτητα δεν επαρκεί όμως. Μπορεί να συνεχίσει κανείς ε, μια πορεία. Αν συνεχίσει όμως την λαθασμένη πορεία μπορεί να βρεθεί είσαι στο έδαφος. Το παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο σήμερα θα κρίνει το τέταρτο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας σε 12 μήνες. Η πλειοψηφία των βουλευτών θα ψηφίσει αυτό το έγγραφο λόγω του περιεχομένου, αλλά και επειδή πρώτα παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες και δεν είχε συζητηθεί ή δεν ήταν γνωστό ή δεν είχε εγκριθεί προηγούμενα στην Πορτογαλία. Γι' αυτό θέτω ένα ερώτημα στην Ουγγρική Προεδρία. Σύμφωνα με τις προθέσεις της θέλει να υπερασπιστεί τον υποχρεωτικό χαρακτήρα αυτών των εγγράφων. Δεν πρέπει αυτές, αυτά τα έγγραφα να έχουν προηγούμενη κοινοβουλευτική έγκριση ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Αύριο το Συμβούλιο θα αποφασίσει για ένα μηχανισμό που θα ισχύει μετά το 2013. Αλλά δεν λέγεται τίποτα για τον μηχανισμό ε, χρηματοδότησης, τον υφιστάμενο που μας ενδιαφέρει. Όταν ε, πέρασε η Πορτογαλία σε αυτό το κύκλο ήταν ε, αναπόφευτη η έκρηξη του χρέους. Και τι έγινε εδώ για την ε, αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας για το χρέος της Πορτογαλίας και να μην μας πούν ότι το θέμα είναι πορτογαλική υπόθεση. Διότι οι ε, περικοπές και οι περιστολέ είναι δικές μας, όμως οι ευθύνε είναι δικέ. σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρντ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων η ΥΠΑΤΟΣ εκπρόσωπος χθε ανέφερε ότι θα υποστηρίξει τη νέα, το, το νέο καθεστώς όσον αφορά και την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών στέγασης δεδομένης της μεγάλης ανέχειας και της φτώχειας που αντιμετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Αιγύπτου δεν μπορεί κανείς να διαφωνεί. Είναι ένα καλό παράδειγμα αλληλεγγύης από βράση της Ευρώπης. Είμαι υπέρ του να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών της Αιγύπτου. Ιδιαίτερα μια και η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο τώρα μετά την αποχώρηση του Πρόεδρου Μουμπάρακα και υπάρχουν, ε, υπάρχει ε, μεγάλη ανάγκη για την ε, διασφάλιση αυτών των πτυχών και των τροφίμων. Εδώ πρέπει να βοηθηθεί αυτή η Νέα Αίγυπτος. Η Νέα Αίγυπτος που άσχετα από την θρησκεία τους οι πολίτες θα είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και θα έχουν ίσα δικαιώματα και η συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ θα πρέπει να είναι σεβαστή και να εφαρμοστεί είναι σημαντικό αυτό και για την εσωτερική και την εξωτερική σταθερότητα της Νέας Αιγύπτου. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά παρακαλώ. <laughs> Eh. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προηγούμενα όμως ε, δεν με είδατε, γι' αυτό σας ευχαριστώ παρόλα αυτά που μου δίνετε τον λόγο και μπορώ να πω και εγώ κάτι. Κυρία Πρόεδρε, θα έχουμε ένα μηχανισμό σταθεροποίησης, ε, ένα ταμείο ε, υποστήριξης ε, που θα μπορεί να δράσει. Αποδέκτες θα είναι άτομα τα οποία έχουν τύχει πολλών δώρων που διαρκώς τις υποσχέσεις τους δεν τις στηρούσαν. Αριθμητικά μεγέθη είχαν νοθευθεί εδώ και χρόνια. Εδώ και δέκα χρόνια για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δινόντουσαν υποσχέσεις ότι όλοι θα τις στηρούσαν, Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα δεν τήρησαν τι υποσχέσει του. Τα μεγάλα ελλείμματα και το χρέο δεν αντιμετωπίστηκαν. Και τώρα δίνονται πάλι υποσχέσει ότι αυτό το σύμφωνο λέει θα λειτουργήσει. Οι ε, Βρυξέλλες καθορίζουν πόσα θα κερδίζει ο μισθωτό στην Ολλανδία. Τι θα παίρνει όσον αφορά τη σύνταξή του. Θα τα πληρώσουν όλα δηλαδή οι πολίτε, οι φορολογούμενοι, στου οποίου δεν γίνονται δώρα. Είναι ένα πολύ ακριβό, δαπανηρό παιχνίδι για τη σελίδα αυτό. Δεν αξίζουν αυτές οι χώρες ε, την εμπιστοσύνη που χρειάζεται το νόμισμα. Υπάρχουν χώρες που δεν τηρούν εντάξει τα οικονομικά τους και τα δημοσιονομικά τους. Αυτές οι χώρες πρέπει να αποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσει το σύμφωνο σταθερό. λόγω του που έκανα, θα είχατε πάντα την ευκαιρία να τα πείτε. Ο κύριος Μάουρο τώρα για δύο λεπτά. Μάουρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε οι αναταραχές που πολλαπλασιάζονται στη Νότια Μεσόγειο δεν θα πρέπει να αποσπούν την προσοχή μας από τους στόχους και οικονομικού χαρακτήρα που από καιρό έχουμε καθορίσει για μεσοπρόθεσμα. Οι διεθνείς αναταραχές θα πρέπει να επιταχύνουν αντίθετα το βήμα για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και είναι καλό οι αποφάσεις για την εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 να εφαρμοστούν γρήγορα κατά τη διάρκεια τη συνεδρία αυτή τη εβδομάδα να ληφθούν οι αποφάσει. Εμεί δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά την σύγκρουση στη Λιβύη, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα είναι όπω πριν. Η Ευρώπη έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να έχει ένα πακέτο μέτρων που θα επιτρέψουν στι οικονομίε των κρατών μελών να ξαναπάρουν ανάσα εν ώψη μια νέα περίοδου αβεβαιοτήτων. Σίγουρα, βεβαίω, το μεγαλύτερο ερωτηματικό συνδέεται με την κατάσταση στη Μεσόγειο. Η Μεσόγειο στον πόλεμο είναι η χειρότερη καταστροφή που μπορεί να περιμένει ε, ο κόσμος σήμερα. Ε, καλά έκαναν οι χώρες που θεώρησαν απαραίτητο να κινηθούν σε αυτή την περίσταση. Κάναν καλά. Παραμένει όμως μεγάλη αντίφαση. Ευρωπαϊκή Ένωση που φαίνεται ε, διαιρεμένη και αναποφάσιστη στο τι θα πρέπει να κάνει και τι θέλει να κάνει. Θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση λοιπόν προς την Ουγγρική Προεδρία. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κοντά σε αυτή την Προεδρία που πρέπει να μεταμορφώσει αυτή την κρίση σε κάτι που δεν επιλύει μόνο ε, τα πράγματα βάζοντας σε κρίση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να μεταμορφώσουμε την υπάρχουσα κρίση σε ευκαιρία για να παράγουμε, να αφήσουμε να γεννηθεί επιτέλους, να ζήσει μια εξωτερική πολιτική που να αξίζει το όνομά της. Με τις ευθύνες μας Έχουμε τις αμφιβολίες μας, έχουμε τα σφάλματά μας και είμαστε τις παραμονές κοσμοϊστορικών γεγονότων και θα πρέπει να επομιστούμε αυτή την ευθύνη μέχρι τέλους, φροντίζοντας ούτως ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν από το Συμβούλιο αύριο και μεθαύριο να μπορούν να είναι λογικές, αλλά πάνω απ' όλα να μπορούν να είναι γενναίες λέει. Ευχαριστώ. Η κυρία για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήδη εδώ αναφέρθηκε ότι δυστυχώς αυτή τη χρονική στιγμή στην Πορτογαλία το ε, Κοινοβούλιο μπορεί να ε, καταρρύψει την κυβέρνηση. Αν ε, ανατραπεί η κυβέρνηση θα υπάρξει αστάθεια πολιτική που θα έχει προκληθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δεν υποστήριξαν άλλο ένα πακέτο μέτρων αυστηρότητας, δημοσιονομικής λιτότητας. Και αυτό όχι επειδή τα προηγούμενα πακέτα δεν υλοποιήθηκαν, υλοποιήθηκαν, αλλά επειδή οι όροι που επιβάλλονται επιδεινώνουν την όρεξη των αγορών και τα θέματα τα δημοσιονομικά και η κατάσταση δημοσιονομική από τον Ιανουάριο τον Φεβρουάριο είχε ένα πλεόνασμα η Πορτογαλία σε σχέση με το 10% και αυξήθηκε, αυξήθηκαν τα έσοδα 11 συνολικά Οι πολιτικές ομάδες που δημιούργησαν αυτή την πολιτική κρίση απορρίπτοντας αυτό το πρόγραμμα λιτότητας που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση και που υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτές οι δυνάμει μπορεί να είναι πολύ ικανοποιημένε με αυτή την κατάσταση. Όμως η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι δημιουργούνται προβλήματα λόγω της υπερχρέωσης και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Είναι το χειρότερο για την Πορτογαλία και για τους πολίτες και για άλλη μία φορά για το θέμα της αηφορίας του μεγάλου εγχειρήματο του κοινού νομίσματος. Δεν βρισκόμαστε σε μια κρίση της ζώνης ευρώ, βρισκόμαστε μέσα σε μια πάρα πολύ σημαντική κρίση της ίδιας, του ίδιου του ευρώ. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους Ποια είναι η εναλλακτική λύση κύριε. Όλα τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα δικά του σχέδια λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας μέχρι τον Απρίλιο. Η Πορτογαλία χρειάζεται περισσότερα μέτρα αλητότητα για να μειωθεί το έλλειμμα και να αντιμετωπιστεί το δημόσιο χρέο. Να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα μέχρι το 2012-2013 και να έχει φτάσει στο 2 3%. Και εδώ δεν υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ λύσει. Το να απορρίπτει κανεί αυτέ τι προτάσει είναι πρόβλημα. Και εδώ ευχαριστούμε για την προσπάθεια των Πορτογάλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντεσάρνες. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο Συμβούλιο έχει την τελευταία ευκαιρία για τους ευρωπαϊκούς ε, ηθήνοντες να ε, μπορέσουν να δράσουν από κοινού εργαζόμενοι στις κοινέ αξίες. Όταν ένας ε, πληθυσμός βάλεται θα πρέπει να προστατευτεί χάρη της Γαλλία έχει λανθεί δράση. Μπορέσαμε να εμποδίσουμε ο Καντάφη να φτάσει στην Βεγγάση. Ωστόσο το, συμβούλιο, το συμβούλιο θα πρέπει να αναγνωρίσει την λιβική αντίσταση για να την ενισχύσει και να απομονώσει περισσότερο τον Καντάφη ούτω ώστε να πέσει επιτέλους αυτή η κυβέρνηση. Και επίσης είναι θεμελιώδες αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μπαχρέν, στη Συρία, στην Ιεμένη και πράγματι είναι πολύ ουσιαστικό αυτό που βλέπουμε, τον κύκλο δηλαδή της βίας να αναφλέγεται στην Μέση Ανατολή. Αναμένουμε από τους ευρωβουλευτές να δράσουν πριν είναι πολύ αργά. Η ιστορία κινείται σε ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου και το πολιτικό σθένος έγκυται ακριβώς στο να σταθεί κανείς ε, αντάξιος αυτών των περιστάσεων και να φτάσει έγκαιρα στο ραντεβού. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το να δίνουμε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ εκ μέρους της Ολλανδίας για εγγυήσεις είναι ο δρόμος προς δημοσιονομικό ή κόλαση μέσω εγγύησεων. Οι εγγυήσει που έχουν δοθεί είναι πάρα πολύ υψηλέ και πάρα πολύ ε, μεγάλο είναι ο κίνδυνο. Δεν ξεπεραστεί με αυτόν τον τρόπο η κρίση διότι τελικά δεν πετυχαίνουν το στόχο. Η κρίση δημιουργήθηκε από ανεύθυνη συσσόρευση χρέους και όχι με τη συμμόρφωση συμφωνιών που είχαν συναθεί. Και αν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, ως εγγύσεις και να δίνουμε δεν θα βοηθήσουν. Θα έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και το 2004 ε, το αγνόησαν και η Γαλλία και η Γερμανία. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να προωθήσουμε αυτό το μέτρο με αυτόματες κυρώσεις τι συμβαίνει με τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Οι κυρώσεις παίρνουν δεύτερη θέση έναντι των πολιτικών συμφερόντων. Τι βλέπουμε, ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν την κατάσταση με, με κινησμό. Αισθάνονται κινησμό. Δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ. Ένα Κυρία Ήλια έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι απαράδεκτο η οδός που ε, πορεύονται οι υπεύθυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την εκμετάλλευση των εργαζομένων με νέα μέτρα αντικοινωνικά που επιδεινώνουν τις ανισότητες αυξάνουν την ανεργία και την ανέχεια της εργασίας την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό πάντα εξυπηρετώντας ε, δυνάμεις μεγάλες ε, οικονομικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το πλούτι τους αυξάνονται διαρκώς και εδώ θέλουν να επιβάλλουν στραγγαλισμό στις πιο αδύναμες οικονομίες και να γίνουν προτεκτοράτα κυρίαρχα κράτη με τους όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζουν για την εφαρμογή όπως λέγεται, όπως από τον αποκαλούν του μηχανισμού σταθερότητας. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σε αυτά τα μέτρα όπως συνέβη το προηγούμενο Σάββατο στην Πορτογαλία στην διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 300.000 άτομα και σήμερα στο, Πορτογα το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας όπου η πλειοψηφία των βουλευτών θα κάνει το ίδιο. Θα καταψηφίσει το τέταρτο πακέτο λιτότητας. Αναφέρθηκε εδώ Πρόεδρε να πούμε όχι στις, ε, στους βομβαρδισμούς ε, που κάνει η Διεθνή Συμμαχία στη Λιβύη και λέμε όχι στην καταπίεση των λαών σε όλους τους λαούς της περιοχής ε, τη Λιβύη, τον Μπαχρέν και την Ιεμένη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Φιγερέδο 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση είναι προαπαιτούμενο για τη σωστή, σταθερή, εύρυθμη λειτουργία νοικοκυριών, επιχειρήσεων, χωρών και μιας ενώσεως χωρών. Βεβαίως, αν μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποφασίσει να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει ένα νέο νόμισμα, πρέπει να υπάρχει και ένας μηχανισμός, ούτω ώστε να αποφεύγεται το γεγονός οι ανεύθυνοι πολιτικοί να υπονομεύουν αυτό το νέο νόμισμα. Και πώς, μέσω δράσεων ε, ψηφοθυρικών. Οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να πληρούν, να συμμορφώνονται με κάποια κριτήρια και κανόνες. Οι κανόνες θεσπίστηκαν με καλούς, ε, καλές προθέσεις αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. είμαι υπέρ αυτομάτων κυρώσεων εάν δεν γίνονται σεβαστοί οι συμπεφωνημένοι κανόνες. Οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο εμπορίας και παζαρέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε συνάδελφε. Δύο λεπτά στη συνέχεια ο κύριος Σάριους Βόλσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω τη γέννηση του, ε, ε του προγράμματος ε, Europlus, που είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Το νέο πακέτο δημιουργείται μια νέα αρχιτεκτονική, περίπου, ε, και αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να είναι πλήρες και ανοιχτό για εκείνους που θέλουν να συμμετάσχουν στο σύμφωνο αυτό για το ευρώ και να μην δημιουργηθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Ε, δυστυχώς το σύμφωνο θα είναι μισό ανοιχτό, διότι η τροπολογία του άρθρου 136 που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ε, κατέπεσε και έλεγε ζητεί ο, στα, στο, ο μηχανισμό σταθερότητα να είναι ευθύς εξ αρχής ανοιχτό σε κράτη-μέλη που δεν έχουν σαν νόμισμα το ευρώ αλλά θέλουν να συμμετάσχουν στο ευρώ θα είναι μισάνοιχτο ο μηχανισμό, διότι θα πρέπει να υπομειστεί υποχρεώσει. δεν θα είναι ανοιχτό ο μηχανισμό για αυτού που είναι εκτό ευρώ και θέλουν να συμμετάσχουν στι τάξει εκείνων που είναι μέσα. Αυτό που μα ενώνει είναι μια αγορά περισσότερο από το ευρώ. Δεν είναι η κρίση στο ευρώ αυτή, αλλά είναι κρίση κάποιων χωρών τη ευρωζώνης και οποιοδήποτε άλλο κράτο που δεν ανήκει στην ευρωζώνη μπορεί να έχει τέτοιο πρόβλημα δημοσιονομικά. Βλέπω έλλειψη λογική και έλλειψη συνέπειας. Ε, κάποια λόγια για την Νότια Μεσόγειο και τη Λιβύη τώρα. Πρώτα απ' όλα, συγχαίρω εμάς, όχι την Ένωση, αλλά κάποια κράτη-μέλη που είναι στην πρώτη γραμμή της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Λιβύη και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς τη Γαλλία και την Ιταλία και προς τον Νίκολα Σαρκοζή που ηγήθηκαν τις προσπάθειες. Νομίζω ότι είναι η απαρχή αλλαγή τη εξωτερική πολιτική. Από εκεί που εκινεί το βάση συμφερόντα να κινηθεί βάση αξιών. Χρειαζόμαστε δύο επόμενα βήματα. Να επανασχεδιάσουμε την πολιτική γυτνίαση και να απευθυνθούμε και προ κοινωνίε, τι κοινωνίε και όχι κυβερνήσει και να κάνουμε μετάβαση ή μεταρρύθμιση, όπω την αποκαλούμε στην κεντρική Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα συναγερμό για μεταρρύθμιση και ενίσχυση τη ΚΕΠΑ να έχουμε δυνατότητες ε, κοινέ στην Ευρώπη για στρατηγικής και ελέγχου των προσπαθειών. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Για τρία λεπτά στη συνέχεια ο συνάδελφος Χουάν Μποκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αύριο στις 24 Μαρτίου θα είναι μια μέρα συμβολικού χαρακτήρα. Καταρχήν θα σηματοδοθεί από την τροποποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας που έχουμε ψηφίσει ούτως ώστε να επιτραπεί η εγκαθίδρυση ενό ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητα, μόνιμου μηχανισμού. Αυτό ο μηχανισμό παρέχει δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, υπάρξουν κάποια ευρωομόλογα ε, ως άμυνα κατά των επιθέσεων των κερδοσκόπων. Ε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε στα μισά του δρόμου. Ε, η αναθεώρηση της συνθήκης θα είναι μια ευκαιρία να δοθεί η άδεια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επαναγοράσει το δημόσιο χρέος, ε, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συσταθεί και το σύμφωνο του ευρώ που δεν είναι τίποτα άλλο από το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Αυτό το σύμφωνο το πρασπίζεται ε, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζετε την ε, συνένεση της ε, Washington. Στις 24 Μαρτίου έχουμε την γέννηση της συνένεσης των Βρυξελών. Η συνένεση των Βρυξελών συνιστά την βάναση εφαρμογή του νεοφιλελεύθερου δόγματος όσον αφορά το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες ε, παροχές θα περικοπούν, θα υπάρχει ελάχιστη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Επιτροπή έχουν βραχυπρόθεσμη μνήμη. Μας προτείνουν να μετασχηματίσουν το σύμφωνο για, την, ε, για το ευρώ στο ε, κάτι που ήταν στην επαρχή της κρίσης. Στην Ισπανία και στις ε, χώρες η άνοδος του χρέους δεν έχει άλλες αιτίε από την κρίση της αγοραστικής δύναμης λόγω της αλλαγής των, και της μίας των μισθών. Το σύμφωνο για το ευρώ προτείνει δυστυχώς να διανυστεί αυτή η λιτότητα στους μισθούς. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, εκτός από το ότι είναι η συνέπεια της κρίσης, είναι επίσης η συνέπεια μιας άχρηστης μίας των επιτοκίων, όπως λένε οι νεοφιλελεύθεροι. Η λιτότητα των μισθών και του προπολογισμού σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, όπως έχει προγραμματιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα καταλήξει να σκοτώσει την ευρωπαϊκή ε, ζήτηση και να σκοτώσει την ανάκαμψη χωρίς να μειώσει το έλλειμμα. Αύριο θα είμαστε στο πλευρό των μισθωτών οι οποίοι θα διαδηλώσουν έναντι αυτής της των Βρυξελών είναι το τρίτο σύμβολο αυτής της ε, ημέρας της 24 η Μαρτίου. Εάν δεν θέλουμε να ανέλθουν οι φαίες, οι συντηρητικές δυνάμεις, η Ευρώπη θα πρέπει να οικοδομηθεί από κοινού με τους ε, λαούς. Ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Γέτεν Μέκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού για τη διαχείριση των κρίσεων για την Ευρώπη είναι κάτι απαραίτητο για να προστατευτούμε από μελλοντικέ κρίσει. Κανεί δεν θέλει μια νέα κρίση, αλλά ίσω τελικά να αντιμετωπίσουμε μια. Είναι ατυχέ το ότι αυτό ο μόνιμο μηχανισμό διαχείριση των κρίσεων έχει σχεδιαστεί εκτό των θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ο μηχανισμός θα έπρεπε να πλησιάσει δυνατόν περισσότερο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση του. Και κυρώσεις θα έπρεπε να είναι αυτόματες και δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και παζαρεμάτων. Και τώρα μερικά λόγια για την εξωτερική πολιτική όπως αποκαλείται της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τη Λιβύη. Η κατάσταση στη Λιβύη ε, είναι συγκεχημένη και έχει προκληθεί και σύγχυση και στη διεθνή κοινότητα. Μία ζώνη απαγορεύσεως των πτήσεων δημιουργήθηκε για να προστατευτούν οι πολίτες και εκεί είχε αναμειχθεί, ε, έχει αναμειχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα που δέχτηκαν επίθεση χερσαίες δυνάμεις θα πρέπει να διαρωτηθούμε κατά πόσο αυτό ήταν ο στόχος της δημιουργίας τόσο απαγορεύσεων πτήσεων. Ίσως τελικά να προωθήσαμε σε άλλο σημείο το καθόφλι του πολέμου. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριο Έπινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπε και ο Σούλτ ότι οι στατικέ επιχειρήσει δημιουργήθηκαν, προγραμματίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Αντιθέτω, ήρθαν πολύ αργά. Η Δύση περίμενε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να απομονώσει στην Τρίπολη τον Κατάφη και να τον υποχρεώσουν να φύγει ή αλλιώ να τον εξαλείψουν. Ε, τώρα ήμασταν ε, μόνο έγκαιροι για να προλάβουμε μαζική δολοφονία στην ε, Βενγάζη. Και βλέπουμε τη Γαλλία και τη Βρετανία οι οποίε ηγήθηκαν. Συγχαρητήρια λοιπόν. Η Γερμανία είναι μια χώρα όπου είναι για το σκληρό νόμισμα και ήπια ισχύ. Ο Υπουργό Άμυνα ε, τελικά στη Γερμανία είναι πιο επικίνδυνη δουλειά. Η Τουρκία είναι εναντίον του ΝΑΤΟ. Και η είναι η χώρα που υποχωρεί, σαν θεατή δρά. Φοβούμαι ότι όπως και στα Βαλκάνια τώρα δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό, αυτή την αποτελμάτωση χωρίς να έχουμε μια συγκεκριμένη αμερικανική ηγεσία. Χωρί αυτή δεν πάει κινηθεί η Ευρώπη. Ο μόνο πολιτικό που ήξερε πώ να αντιμετωπίσει τον Καντάφη, κύριε Πρόεδρε, ήταν ο Ρόναλντ Ρέγκαν. Ο Ρέγκαν είχε δίκιο πάντα από τότε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε. Για ένα λεπτό στη συνέχεια ο κύριος Χουντής. Κύριε συνάδελφοι, πριν ένα ακριβώς χρόνο η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Έλληνας Πρωθυπουργό αποφάσισαν η Ελλάδα να παίξει το ρόλο του κοινωνικού και του οικονομικού πειραματόζωου. ελήφθησαν λοιπόν ακραία αντικοινωνικά μέτρα με πρόσχημα τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους και της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας. τα αποτελέσματα το χρέος πλησιάζει το 150%, δεύτερο η ανεργία είναι στο 15%, η ανεργία των νέων στο 30%, ο πληθωρισμός στο 4,4%, η ύφεση στο μείον 6,6% στο τελευταίο τετράμινο του 2010. Κύριε Ρεν, το πείραμα το ελληνικό απέτυχε, το πειραματόζω είναι έτοιμο να το εξοντώσετε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ίδιο, την ίδια μοίρα επιφυλάσσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα άλλα κράτη με το σύμφωνο για το ευρώ, δηλαδή την ελληνική την ευρωπαϊκή εκδοχή του ελληνικού μνημονίου είμαστε εναντίον αυτού του συμφώνου διότι δεν θέλουμε την εξόντωση των εργαζομένων των συνταξιούχων και των ανέργων. κύριε Ερέν, όταν υπεγράφει το ελληνικό μνημόνιο ευχηθήκατε στους έλληνες καλό κουράγιο. αν είσαστε συνεπείς στις ευχές την παρασκευή το σάββατο πρέπει να πείτε το ίδιο καλό κουράγιο και στους ευρωπαίους εργαζόμενους. ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Για δύο λεπτά στη συνέχεια ο πρόεδρος μας Hans Gerd αξιότιμε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πολιτιολόγος Αμερικανός Σάμιορ Χάντινγκτον ε, είχε προαναγγείλει τη σύγκρουση των πολιτισμών Clash of, of Civilizations. Αν τον είχαμε πιστέψει θα ήταν μια προφητεία που θα είχε υλοποιηθεί. Εμείς όμως ως Ευρωκοινοβούλιο ε, στοιχηματίσαμε στη συνεργασία με τα αραβικά κράτη και τους ανθρώπους των αραβικών κρατών. Και τώρα βλέπουμε στον αραβικό κόσμο που προσπαθούν να υπερασπιστούν αξίες που και εμείς ε, τις υπερασπιζόμαστε. Την δημοκρατία, την ελευθερία, κράτος δικαίου. Πριν από κάποιες εβδομάδες ποιος θα ανέμενε ότι ο αραβικός σύνδεσμος σε εμάς ε, την δυτική κοινότητα, την διεθνή κοινότητα κρατών θα ζητούσε να σταματήσει η πορεία, να σταματηθεί η πορεία του τυράννου της Λιβύης. Είναι δραματικές αλλαγές αυτές και δεν πρέπει να κάνουμε σφάλματα τώρα. Δεν επιτρέπεται μόνο στα λόγια να βρισκόμαστε στο πλευρό των αραβικών κρατών και των Αράβων. Πρέπει με, με πράξεις που θα ακολουθήσουν τα λόγια να δραστηριοποιηθούμε. Για το Ίδρυμα Κόνραντ Άντεναουερ που είμαι πρόεδρος αυτού του Ιδρύματος θα πάω στην Τινησία. Πριν δύο εβδομάδες ήμουνα στο Κάιρο και θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είπε ο Κόνραντ Άντεναουερ, πρώτος καγκελάριος μετά την, ε, τον πόλεμο της ε, Γερμανίας. Είμαστε στο πλευρό της ελευθερίας, υποστηρίζουμε την ελευθερία. Και εμείς πρέπει να πούμε στους Άραβες, αν θέλετε κι εσείς το ίδιο, τότε είμαστε στο πλευρό σας, ε, με συμβουλές, να σας βοηθήσουμε να προπαρασκευάσετε τις εκλογές, την ελευθερία σας. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ακούμε τώρα ότι στην Ιερουσαλήμ υπήρξε μια τρομοκρατική απόπειρα. Πολλά θύματα θύματα υπήρξαν, πολλοί τραυματίστηκαν. Καταδικάζουμε αυτούς τους ε, ε, υπεύθυνου αυτής της τρομοκρατικής πράξης, όποιοι και να είναι. Πρέπει όμως να υπάρξει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Όταν υπάρχει ο άνεμος της ελευθερίας που φυσά στα κράτη αυτά τα αραβικά κράτη. Πρέπει επιτέλους να υπάρξει ειρήνευση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Να ζήσουν οι Ισραηλινοί μέσα σε ένα ειρηνικό καθεστώς αλλά και οι Παλαιστίνοι να ζήσουν σε ασφαλή σύνορα με αξιοπρέπεια. Αυτός, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να συνεισφέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον αραβικό κόσμο να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Ευχαριστώ. Gracias. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ συνάδελφε Πέτερινγκ. Για δύο λεπτά στη συνέχεια ο κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέρα από τα μέτρα τα οποία προαναγγέλθηκαν, διερωτώ με αν ο ρόλος της ευρωπαϊκής πολιτικής είναι σήμερα στο ύψος των περιστάσεων. Σίγουρα για να επιβεβαιώσει κανείς πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξωτερική πολιτική χρειάζεται αναγκαίος χρόνος αλλά όπως γνωρίζουμε υπάρχουν καταστάσεις όπου διαμορφώνονται και δεν αφήνουν χρονικό περιθώριο αυτό που θέλουμε. Αντίθετα απαιτούν ταχύτητα και μακρόπνοη θεώρηση των πραγμάτων. Σε αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο και κυρίως στη Λιβύη ε, είμαστε υπολοιπόμεθα των απαιτήσεων. Χρειάζεται κάποιος προβληματισμός παραπάνω και να αναγνωρίσουμε ότι ενδεχομένως χρειαζόμασταν μια πρωτοβουλία πιο ισχυρή. Και για να καταλάβουμε τι συνέβαινε, και για να θέσουμε επιτόπου συντονισμένη δράση προς την Μεσόγειο. Δεν μας διαφεύγει, διαφεύγει κανένας ότι αν κοιτάξουμε προς τη Λιβύη βλέπουμε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ της δράσης της κοινής όλης της Ευρώπης και μιας δράσης των, ε, πιο, των κρατών που είναι πιο δραστήρια όπως τώρα. Και το λέω αυτό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποιε ερωτήσει όπου το Συμβούλιο δεν έδωσε απαντήσει και πρέπει να τι δώσει γρήγορα τι απαντήσει. Διερωτώ με αν πέρα από την ανθρωπιστική προσπάθεια έχουμε επίγνωση του τι πρέπει να κάνουμε αν η εφαρμογή του ψηφίσματο 1973 δεν θα αρκεί και αν κάποια χώρα ξεπεράσει τα όρια τη εντολή. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζω την άποψη του Συμβουλίου του θέματος ε, το, της ηγεσία της αποστολής. το ΝΑΤΟ λέει ότι παίζει ρόλο επιχειρησιακό. Χρειάζεται ίσως πιο ενωτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να μην το αναθέτουμε σε κάποιον που είναι πρόθυμος να το κάνει, να το κάνουμε εμείς. Το πλαίσιο των επιχειρήσεων και οι σχέσει με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο και την Αφρικανική Ένωση είναι ουσιαστική σημασία, ούτω ώστε η παρέμβαση στο τέλο να μην θεωρηθεί ότι είναι κάτι αρνητικό και ίσως να δημιουργήσει ε, κινδύνους και άγνωστες παρέκκλησης. Υπάρχει αυτή η επίγνωση. Ίσως δεν υπάρχει στο σύνολό της. Ίσως αυτά τα ερωτηματικά χρειάζονται απαντήσεις πολιτικές επαρκής και όχι γραφειοκρατικές απαντήσεις. Και ξεκινώντας από το αυριανό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε συνάδελφε για ένα λεπτό κύριος Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι σε σχέση με τις ε, κριτικές που ακούγονται ότι δείχνει η Ελλάδα ότι δεν λειτουργεί το ευρώ, είναι καλύτερο να βρίσκεται εκτός ε, συνεργασίας. Όμως αυτοί που λένε αυτά δεν έχουν δίκιο. Η συνεργασία έχει δημιουργήσει σταθερότητα, χαμηλό πληθωρισμό και πάρα πολλές νέες θέσεις απασχόλησης και ο μόνιμος μηχανισμός ε, για την κρίση θα λειτουργήσει ως ε, ίστατη λύση όταν μια χώρα θα έχει τεράστια προβλήματα για τα αίτια της κρίσης αυτά δεν μπορούν να αποφευθούν. Όμως μπορούμε να μεριμνήσουμε το κοινό νόμισμα να είναι ένα σημαντικό μέρος της εξίσωσης της λύσης και να διασφαλίσουμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, λυπούμε για το ότι στη Σουηδική Ράιξτακ, τη Σουηδική Βουλή δεν υπάρχει πλειοψηφία ώστε η Σουηδία να συμμετάσχει στο σύμφωνο του ευρώ. Αυτό σίγουρα μειώνει την επιρροή της χώρας μου Τώρα η Σουηδία αν θα ήθελε να ανήκει στον εσωτερικό πυρήνα του ευρώ τότε δεν μπορεί να παραμένει κανείς εκτός του κοινού νομίσματος όπως και άλλοι αυτά τα οποία λένε πρέπει να ακολουθούνται από πράξεις. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό στη συνέχεια ο συνάδελφος ΣΑΣ Παρακαλώ. Η καταδικάζει το νέο υπεραλιστικό παράνομο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία, η Βρετανία και το ΝΑΤΟ ενάντια στη Λιβύη. Αποτελεί επέσχυντη υποκρισία του ενδιαφέρον για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ο πραγματικός στόχος των υπεριαλιστών είναι τα πετρέλαια το φυσικό αέριο οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της λιβύης της βόρειας αφρικής και της ευρύτερης περιοχής. η υπεριαλιστική επιθετικότητα η νατο και ευρωπαϊκής ένωσης αυξάνει του κινδύνους σε βάρος των λαών της ευρύτερης περιοχής. το νέο σύμφωνο και η ευρωνοσιακή οικονομική διακυβέρνηση φέρνουν μαζική ανεργία φτώχεια ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης αποτελεί μηχανισμό ελεγχόμενης πτώχευσης και σίγουρης χρεοκοπίας για τους λαούς για να προστατευτούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας. αυτός είναι ο ελεύθερος κόσμος των ηπα. αυτή είναι η ευρωπαϊκή ένωση της δημοκρατίας και ελευθερίας. το πραγματικό δίλημα που τίθεται είναι το εξής θα πτωχεύσει ο λαός ή η πλουτοκρατία. για να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες της υπεριαλιστικής βαρβαρότητας και της καπιταλιστικής κρίσης για να μην καταδικαστεί μόνιμα στην ανεργία και τη φτώχεια καλούμε τους λαούς να ξεσηκωθούν ενάντια στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις για να αντεπαιδευθούν για να παλέψουν για τα σύγχρονα δικαιώματά τους για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων. Ευχαριστούμε πολύ συνάδελφοι. Για δύο, λόγο, για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Ράγγελ, ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επισήσω την προσοχή σας για την αξία που δίνει το ΕΛΚ και ιδιαίτερα εμείς οι Πορτογάλοι του ΕΛΚ που δίνουμε στο επόμενο Συμβούλιο για να εξευρεθεί η λύση αυτή που ε, αναμενόταν και για τη δουλειά των ε, συναδέλφων Μπροκ και Γουαλτιέρη που προετοίμασαν τη γνωμοδότηση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί εδώ ο πυρήνας της κοινοτικής λύσης και να μπορέσουμε να αποφύγουμε την διακυβερνητική προσέγγιση. Θα ήθελα να πω στους συναδέφους, αυτή τη στιγμή ζει μια κρίση η Πορτογαλία και το πέστε ε, όσον αφορά την προετοιμασία των εκλογών για να αναλάβει τα ενία της χώρας, να κυβερνήσει τη χώρα σύμφωνα με τα κριτήρια, τα κριτήρια της ζώνης ευρώ, να υλοποιήσει όλες τις προκλήσεις και τα ορόσημα και πέρα από αυτό να κάνει εκείνο που κατά τη διάρκεια 13 ετών το Σοσιαλιστικό Κόμμα 13 ολόκληρα χρόνια το Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν ανίκανο να κάνει. Όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν στην Πορτογαλία είχαν προβλεφθεί από το ΠΕΣΔΕ στι ε, προηγούμενε εκλογέ. Εγώ είχα συμμετάσχει σε αυτή την ε, εκλογική εκστρατεία και είχαμε προαναγγείλει το τι θα συνέβαινε και συνέβησαν αυτά. Και θα, δώσουν, θα υπάρξουν όλε οι εγγυήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στου εταίρου τη ζώνη ευρώ, τη υλοποίηση όλων των κριτηρίων που είναι αποφασιστική σημασία και απαιτητικά κριτήρια, αλλά θα μπορέσουμε να δράσουμε και να ε, υπάρξει η ανταπόκριση. Χρειάστηκαν τέσσερα προγράμματα για την σταθερότητα και την ανάπτυξη και που διαρκώς αναζητούν νέες λύσεις χωρίς να είναι σε θέση να δώσουν μια αξιόπιστη απάντηση στις αγορές, χωρίς να δώσουν μια αποτελεσματική απάντηση στα συμφέροντα των Πορτογάλων και τα συμφέροντα της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Υπήρξαν δύο άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ε, σήκωσαν ε, την μπλε καρτέλα. Καταρχήν η κυρία Εστρέλα. Έχετε μισό λεπτό για την ερώτησή σα, κυρία Εστρέλα. Πρόεδρε, μόνο απλά θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο βουλευτή, ευρωβουλευτή Παύλο Ρανζέλ. Δεν είναι νηπιώδε να λέει ότι πληρώνει υπερβολικά, θα πληρώσει υπερβολικά ακριβά η Πορτογαλία και θα υπάρξουν θυσίε για του Πορτογάλου ε, όταν αναφέρεται εδώ ότι η επόμενη, λέει, κυβέρνηση θα υποβάλει ακριβώ τα ίδια μέτρα ε, λιτότητα και πειθαρχία για να πετύχει, λέει, του στόχου που διαπραγματεύτηκαν τις Βρυξέλλες. Θα ήθελα να μου το απαντήσει αυτό. Δεν είναι μόνο η αγωνία να λάβουν την εξουσία που τους κάνει να τα λένε και να τα κάνουν όλα αυτά. Για να απαντήσετε, έχετε μισό λεπτό παρακαλώ στη διάθεσή σας να απαντήσετε. Θα απαντήσω ευχαρίστως παρότι εδώ μετατρέπεται η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα ε, πορτογαλικής πολιτικής. Εδώ υπάρχει μια απλή λύση. Εμείς πρέπει να κάνουμε εκλογές και θα υπάρξει η ευκαιρία σε σχέση με αυτές τις εκλογές ε, να δείτε τι θα αποφασίσουν ε, οι πολίτες και το τι στοχεύει να κάνει το ΠΕΣΔΕ για την Πορτογαλία. Εγώ λέω δεν μπορούμε να αντέξουμε πια άλλο αυτή την κυβέρνηση που απέτυχε τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Είναι απαράδεκτο δεν είναι αξιόπιστο για τι αγορέ και είναι απαράδεκτο για το Σοσιαλιστικό Κόμμα αυτό που συνέβη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ραζέλ. Η κυρία Γιακονσάρη παρακαλώ. Ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα εδώ να πω στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο δεν μπορώ να ρωτήσω, να θέσω την ερώτηση. Γι' αυτό ερωτώ εσάς άμεσα το ΕΛΚ, την πορτογαλική ομάδα του ΕΛΚ. Γιατί δεν υποστηρίζετε αυτή την πρόταση που είναι τόσο σημαντική. Διότι διαφορετικά όλη η Ευρωζώνη θα υπονομευτεί και θα ε, ζήσει μια κρίση αν δεν περάσει αυτή η πρόταση. Θα ήθελα να μου απαντήσετε και να μου πείτε γιατί η ομάδα σας στην Πορτογαλία αντιστέκεται και διαφωνεί. Υπάρχουν δυσκολίες λοιπόν για να ακούσει κανείς τη συνάδελφο. Υπήρξαν δυσκολίες να την παρακολουθήσει κανείς. Μπορείτε να απαντήσετε. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα υποστηρίζει με ευθύνη όπως έγινε από άλλα, από άλλα κόμματα σε άλλες χώρες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης το πακέτο μέτρων λιτότητας. Όταν απέτυχε αυτή η κυβέρνηση και δεν ήταν σε θέση να δείξει ένα αποτέλεσμα θετικό σε δύο ολόκληρα χρόνια, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να βρεθεί στο πλευρό της λύσης. Και η λύση, η μόνη λύση είναι νέες εκλογές, νέα κυβέρνηση, νέα αξιοπιστία για την Πορτογαλία και για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ραζέλ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Μπουσούτη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες αυτό το Κοινοβούλιο θέτησε ένα ψήφισμα το οποίο ήταν ιδιαίτερος γενναίο σε ένα πολιτικό επίπεδο. Κάναμε μια έκκληση για την ε, δημιουργία μιας ζώνης απαγόρευσης των πτήσεων πάνω από τη Λιβύη. Μόνο, ε, πριν από μια εβδομάδα συναντηθήκαμε σε αυτή την αίθουσα και πάλι. Το ψήφισμα δεν είχε ακόμα εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και υπήρξε ε, μια αίσθηση απογοήτευση, απόγνωση αν θέλετε, γιατί ακριβώς προβλέπαμε την αποτυχία και την, και την ε, απώλεια της Φεγγάζης. Τώρα γνωρίζουμε ότι το ψήφισμα έχει εγκριθεί ε, δύο εβδομάδες μετά. Ε, πιστεύω κύριε Πρόεδρε το ψήφισμα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό και θα έπρεπε να συνεχίσει να εφαρμόζεται ούτω όταν μπορέσουμε να παράσουμε αποτελεσματική βοήθεια προς τον λιβικό λαό και να αποτρέψουμε την αιματοχυσία η οποία συνέβη στην Λιβύη και να τους ε, οδηγήσουμε προς το δημοκρατικό δρόμο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παράσχουμε την ανθρωπιστική μας ε, βοήθεια και συνδρομή, ιδιαίτερα προς εκείνους τους ε, πρόσφυγες οι οποίοι διαφεύγουν προς την την Ισία και την Αίγυπτο. Θα θα υπάρξει ενδεχομένως και μία ροή προσφύγων προς τις δικές μας χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή δεν είναι μόνο μία ευθύνη των ε, μελών της Μεσογείου, αλλά όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριε Μπουσούτιλ. Ε, για 1,5 λεπτό ο κύριος ε, Κέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αίθουσα συνεδριάσεων της, ε, του ΕΛΚ ε, ονομάστηκε επίσημα με το όνομα ε, Αλκίδε Γκάσπερι, ενός από τους ιδρυτές πατέρες τη Ένωση. Τότε ήταν υπερεθνική προσέγγιση για την επίλυση των κρίσεων. Πρώτα απ' όλα προστατευόταν τα ευρωπαϊκά κοινά συμφέροντα. Ήταν ανάμεσα σε εκείνου του ηγέτε που έχοντας γεννηθεί το 19ο αιώνα ήταν σε θέση να αναπτύξει ένα όραμα μιας Ευρώπης για τον 21ο αιώνα όσον αφορά τη σημερινή οικονομική κρίση, ε, χρειαζόμαστε εδώ ηγεσία. Έναν ηγέτη που δεν θα λαμβάνει υπόψη του τι θα γίνει σε επόμενες εκλογές και δεν θα πρέπει να συγκεντρώνεται ο ηγέτης επί της εθνικής διάσωσης, αλλά θα λαμβάνει υπόψη του πώς θα διασωθεί η Ευρώπη και επόμενες γενναίες στο σύνολό τους. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλωσορίζω το νέο κείμενο του Μηχανισμού Σταθερότητας και το πακέτο για την μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Δεύτερον, ελπίζω ότι το, το πακέτο ανταγωνιστικότητας και το σχετικό σύμφωνο ε, θα είναι ανταγωνιστικό και θα προσελκύσει και χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Είναι σημαντικό κάθε κυβέρνηση να αναλάβει εθνικές υποχρεώσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσεως της κάθε χώρας. Τρίτον, για την ενιαία αγορά ανησυχώ λίγο. Θεωρώ ότι οι φιλόδοξοι στόχοι του έχουν περικοπεί σημαντικά και οι ελλείψει οι τη εσωτερική αγορά αγοράς ε, ίσως να αποκτήσουν και μεγαλύτερη σημασία. Σχεδιάζοντα λοιπόν νέα βήματα, α αποδείξουμε ότι έχουμε αξιοπιστία πολιτική και βούληση ολοκληρώνοντας τέσσερι ελευθερίε επί των οποίων βασίζεται η συνεργασία στην Ευρώπη συμπεριλαμβανόμενης τη εσωτερική αγορά και τη εφαρμογής, ε, της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας περί υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλαν. 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο Βαντεκάμπα. Ευχαριστώ. πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τη συμπάθειά μου και τα συλληπιτήριά μου προς τον λαό της Ιαπωνίας. Γνωρίζουμε ότι ε, θα έχουμε μια συζήτηση για την Ιαπωνία σε λίγα λεπτά, αλλά ελπίζω ότι τις επόμενες ε, μέρες το Συμβούλιο θα κάνει δεκτό με της ε, Ιαπωνίας για συνδρομή. Εγώ, εδώ πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χώρα η οποία υπέστη μια ε, τρομακτική καταστροφή και χρειάζεται βοήθεια. Τώρα θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της ε, Λιβύας. Λιβύης. Εκφράστηκαν πάρα πολλά ε, για την Λιβύη. Ε, το ίδιο έπραξε και η Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν να, δεν μπορέσαμε να προσεγγίσουμε την ε, κρίση ωστόσο της πόλης της Λιβύης, δεν μπορέσαμε να αναχαιτήσουμε τα στρατεύματα του, τις δυνάμεις του Καντάφη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή τον πρόεδρο Σαρκοζή, ο οποίος φρόντισε η Ευρωπαϊκή Ένωση τελευταία στιγμή να τη κάτι από κοινού με το ΝΑΤΟ. Αλλά δυστυχώς η οδύνη των ανθρώπων παραμένει. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε κάπως ε, σεμνοί. Μετά την κρίση η Ευρώπη ε, ε, είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι πριν. Τώρα, όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητα, εδώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Ο κ. Μπαρόσο το αποκάλεσε ακρογωνιαίο λίθο. Αλλά κατά την άποψή μου όλα αυτά είναι κάπω ε, χαλαρά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δουλέψω σε την κατεύθυνση προσεχή μήνε. Αύριο θα έχουμε απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει 1,5 λεπτό ο κύριος Σκέλης. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στην οικονομική πτυχή, διότι η χώρα μου που είναι αποδέκτης ε, ε χρημάτων Ευρωπαϊκή Ένωση μπορώ να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Έχουμε νέα κυβέρνηση όμω και έχουμε νέα ελπίδα στην Ιρλανδία και η πρώτη ομιλία που έκανε ο πρόεδρό μα, ο Τίσοκ, είπε ότι θέλει να δημιουργήσει γέφυρε στην Ευρώπη ε, και να φέρουμε το βάρο μα τελικά και να επηρεάσουμε την κατάσταση. Με δύο τρόπου πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα το επιτόκιο είναι δρακόντιο και δεν είναι βιώσιμο. Θέλουμε αυτό να μειωθεί κατά τουλάχιστον 1 με 2%. Δεύτερον, χρειαζόμαστε συνεχή εγγύηση χρηματοδοτήσεως των τραπεζών μας ώστε να, λειτουργήσουν ξανά. Δεν χρειαζόμαστε πιέσει όσον αφορά τον φόρο επί των επιχειρήσεων και δεν χρειαζόμαστε διαλέξεις από τύπου σαν τον κύριο Σαρκοζή που φαίνεται να αισθάνεται πολύ άνετα με ένα υψηλό ποσοστό στη Γαλλία Δύο κάτι, ενώ το δικό μας είναι 11,9. Θα έπρεπε να δει τα του οίκου του πριν ρίξει τη μάτια του πέρα από την Ιρλανδική θάλασσα. Λοιπόν, πού, πώς γίνεται, πού υπάρχει το αντάλλαγμα ένα προς ένα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε το, τα μέτρα ε, λιτότητας και θα βοηθήσει αυτούς τους πολίτες μας. Δεύτερον, θα δούμε κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό εφαρμόζει η Γερμανία το 2009 για το χρέος. Τρίτον, Θέλουμε ευρωπαϊκό φορέα ανεξάρτητο οικονομικό φορολογικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι δεν υπάρχει εθνική τέτοια υπηρεσία ανεξάρτητη. Είναι τα γενέθλιά του σήμερα του κ. Μπαρόσο. Και ζητώ από αυτόν και του συναδέλφου να βοηθήσουν και το Κοινοβούλιο να, βοηθήσει, ε, να μας βοηθήσετε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εμείς τον εαυτό μας σαν χώρα και να ζητήσουμε ξανά βοήθεια στο μέλλον. Σα κύριος Λίσεκ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, συνάδελφοι. Είναι καλό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρήκαν τόσο χρόνο τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες να αφιερώσουν την προσοχή τους όσα εκτένονται στη Βόρεια Αφρική και στη Λιβύη και ελπίζω ότι ε, η σφαγή των αμάχων θα μπορέσει να σταματήσει και ότι θα μπορέσουν οι Λίβοι να ανατρέψουν τον τύρανο στην Λιβύη. Όμως υπάρχουν και εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα που συσχετίζονται με την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, με την εξωτερική πολιτική. Υπάρχουν διαφορές απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει πόσο πόρο απέχουμε από τον κοινό στόχο να έχουμε μια πραγματικά κοινή κοινοτική πολιτική και σύμφωνα με τις συνθήκες της Λισαβόνας είναι πρόκληση αυτό για την διεθνή κοινότητα. Καλό είναι ότι συνεργαζόμαστε με τη ΣΥΠΑ και με άλλες χώρες. Καλό είναι ότι έχουμε διάλογο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Αφρικανική Ένωση. Καλό είναι ότι υπάρχει και ο διάλογος με το Ισραήλ. Και όπως ο πρόεδρος Hans Gert Pöttering προανέφερε, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Βόρεια Αφρική, στην Λιβύη, αυτά που συνέβησαν στην Αίγυπτο, θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες επιπτώσεις για την διαδικασία ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής. Να το θυμόμαστε πάντα αυτό θα έπρεπε να προβληματιστούμε για το μέλλον, να σκεφτούμε το μέλλον, να προάγουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι πυροσβεστικά. Θα έπρεπε να σκεφτούμε και για τις άλλες χώρες ε, που βρίσκονται γύρω από τα σύνορα της Ευρώπης και που παρόμοια προβλήματα θα αντιμετωπιζόντουσαν. 1,5 λεπτό κύριος Γκάλερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε στα Ισπανικά. <clears throat> Στο ε, ε, σημείωμα πρόσθεσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει ο κύριος Φανρόμποϊ το γεύμα μας ε, θα το ξεκινήσουμε με μια επισκόπηση της κατάστασης ε, στην Βόρεια Αφρική στη Λιβύη Ελπίζω ότι θα αποσταλούν σαφή μηνύματα και από κοινού θα σταλούν κοινά μηνύματα στον Καντάφη, στους πολίτες της Λιβύης, αλλά και στους δικούς μας πολίτες που έχουν ενοχληθεί για αυτές τις διαφωνίες που υπάρχουν όσον αφορά ε, την απέτηση να βρίσκεται στην εξουσία ένας δικτάτορας. Και θα πρέπει εδώ να ε, υπάρξει η δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Όμως θα επιθυμούσα πέρα από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί του ΝΑΤΟ να θυμόταν τις αποφάσεις της όσον αφορά το δυναμικό και τις δυνατότητες ε, και το ναυτικό των κρατών μελών να είχε επιβάλει τον αποκλεισμό της Λιβύης. Στο κάτω-κάτω δική μας γείτονα είναι η Λιβύη. Και έτσι αυτές οι εντάσεις με την Τουρκία θα είχαν αποφευθεί και θα είχε ανακουφιστεί ε, ο σύμμαχός μας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή η κυβέρνηση. Και τώρα σε σχέση με τους ε, πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ισία και την Αίγυπτο θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε με την ανθρωπιστική βοήθεια να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι απόλυτη ανάγκη. Να δείξουμε στους ε, Λίβιους ποιοι είναι οι στόχοι μας. Και για τους συναδέφους ε, των, ε, του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος μόλις άκουσα ότι πέθανε ο Στάλιν αλλά και έχουν αποσταλεί νέες οδηγίες του Πολίτμπυρο αλλά δεν έχουν φτάσει φαίνεται αυτές οι οδηγίες αυτούς. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος Πρέντα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι ο τελικός στόχος στην παρέμβασή μας αυτή, στην επέμβασή μας στη Λιβύη είναι να πάψουν οι βιοπραγίες και οι απαράδεκτες αυτές ε, ομότητες του καθεστώτος του Γκαντάφη έναντι των εξεγερμένων το ψήφισμα 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών διασφαλίζει το γεγονός ότι εμείς θα μπορούμε να θεσπίσουμε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων για να προστατεύσουμε τους αμάχους. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι πρωτού υιοθετηθεί το ψήφισμα 1973 από το Συμβούλιο Ασφάλειας, το Ευρωκοινοβούλιο ήταν το πρώτο ε, παγκόσμιο θεσμικό όργανο που είχε ζητήσει την θέσπιση μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και είχε ζητηθεί αυτό από το Ευρωκοινοβούλιο στην προηγούμενη είναι Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Νομίζω εδώ υπάρχουν τα εξή στοιχεία για να διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματο στη Λιβύη το κύριο σύνθημα θα πρέπει να είναι συντονισμό και σαφήνεια. Συντονισμό πρώτα και κυρία στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τι ε, διατάξει συνθήκη όσον αφορά και τι ανθρωπιστικέ πτυχέ. Συντονισμό. Συντονισμό όσον αφορά το ΝΑΤΟ. Οι δράσει μα πρέπει να είναι συμπληρωματικέ των δράσεων του ΝΑΤΟ. Χρειάζεται συντονισμό και με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Διότι πρέπει να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τι δυνάμει σε αυτή την περιοχή ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του εγχειρήματό μα στην Λιβύη. Όταν πρόκειται για το σθένος μας να σταματήσουν οι ομότητες κατά των αμάχων, όταν πρόκειται για την καθαρότητα του μηνύματός μας, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να οδηγήσουν στην επιτυχία της δράσης μας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τον γύρο των παρεμβάσεων από τα μέλη, από τους ευρωβουλευτές και περνάμε τώρα, θα δώσουμε τον λόγο σε εκείνους τους συναδέφους που πρόσεξε ο πρόεδρος στη διαδικασία Κάτσιδια. Είναι νέα αυτή. Θα δώσουμε τον λόγο σε όλους, παρότι αυτό ξεπερνά λίγο περισσότερο τον χρόνο από ό,τι επιτρέπει ο κανονισμό. Θα αφαιρέσω τον λόγο αμέσω όταν θα έχει ολοκληρωθεί το ένα λεπτό από αυτού. Πρώτα απ' όλα η κυρία Γκάλπεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Ε, Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, σύμφωνα με τους πρόσφατες οικονομικούς δείκτες βγαίνει η Ευρώπη από την κρίση. Αυτή είναι μια ε, διαδικασία που προωθήσει το επικείμενο Συμβούλιο. Ε, υπήρξε κάποια κίνηση και είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη έφτασε σε νέα επίπεδα. Ένα πακέτο μέτρων εμπεριέχει σημαντικά στοιχεία όπως είναι ο μακροοικονομικός συντονισμός και ο σχετικός κύκλος όπως το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και η Ουγγρική Προεδρία του Συμβουλίου ετοίμασε σχετική συνοπτική έκθεση. Πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον μας μετά την κρίση και τι μπορεί να αναμένεται τότε στο μέλλον. Η Ουγγρική Προεδρία επίσης διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Έγιναν αποδεκτοί γενικοί προσανατολισμοί, εγκρίθηκαν, άρα μπορούμε να δούμε νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ουγγρική Προεδρία για τα όσα έλαβαν ε, την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι μια επιτυχία. Ευρωπαϊκή επιτυχία επίσης αυτή. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε ότι θα δημιουργηθούν οι βάσεις για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και για την δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την οικονομική πολιτική. Αυτό θα είναι ε, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα συνεπάγεται μια νέα φάση. Σε αυτό το νέο πλαίσιο που θα δημιουργήσουμε η ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ θετικό να μπορέσει να εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση αυτό το εγχείρημα, αυτό το πακέτο των έξι ε, μέτρων, νομοθετικών μέτρων. Διότι αν υπάρξει καθυστέρηση όλη η Ευρώπη θα ζημιωθεί συνολικά. Σας ευχαριστώ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ το Συμβούλιο για την ελαστικότητά του και διακόπτεται. Ο κύριος Γκάλαγκερ στη Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ιρλανδική κυβέρνηση για να πετύχει μία μείωση ε, του επιτοκίου όσον αφορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ενώσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε πρόθυμη να υποστηρίξει μία μείωση του επιτοκίου και ελπίζω ότι τα 27 κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να καταλήξουν σε μία συμφωνία όσον αφορά την αναθεώρηση του όλου ζητήματος η Ιρλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το χρέο μα θα είναι βιώσιμο. Είναι ουσιαστικό η τιμολόγηση τη οικονομική βοηθείας και του σχετικού μηχανισμού ε, να είναι κάτι που να μπορεί να το αντέξει κανεί να το πληρώσει και να είναι δίκαιο. Κάποιες χώρες επιδιώκουν εκχωρήσει από την Ιρλανδία με αντάλλαγμα μείωση του επιτοκίου. Και βεβαίω από ό,τι φαίνεται η πίεση επί τη Ιρλανδία υπάρχει να αυξήσει τον φόρο επί των επιχειρήσεων. Δεν έχω χρόνο να επισέλθω ε, σε λεπτομέρειες τι γίνεται με τον άλλο φόρο εκτός του φόρου επί των επιχειρήσεων και εδώ διακόπτεται το μικρόφωνο. Ο κύριος Μπρόντς έχει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, που διέκοψε τον προηγούμενο μιλήτη. So Council... Ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θετήσει την απόφαση για τροποποίηση της συνθήκης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτό υποτίθεται ότι θα κρατήσει, θα βοηθήσει τι χώρε να μείνουν εντό ευρωζώνη. Θα αποτύχει βεβαίω, όχι λόγω ελλείψεω χρημάτων, που ρίχνουν στο πρόβλημα, αλλά γιατί το πρόβλημα είναι ενδημικό. Είναι ένας μηχανισμός που προσπαθήσει να κάνει το νερό να κυλήσει προς την ανηφόρα. Λοιπόν, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται η ζήτηση και η προσφορά για το νόμισμα μιας χώρας και θα πρέπει αυτό να αντικατοπτρίζει την, αίτηση, την ζήτηση για τις εισαγωγές και εξαγωγές της χώρας και ροές κεφαλαίους. Η ίδια αξία του συναλλάγματο δεν μπορεί να αντικατοπτρίσει ε, την οικονομική κατάσταση 17 χωρών. Αντί να υπάρχει ένα μηχανισμό που θα πρέπει να βοηθά τι χώρε που είναι εντός Ευρωζώνης, χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό για να τι σώζουμε από το ευρώ. Ακόμα και οι χώρε αυτέ που είδαν επιτυχίε στην Ευρωζώνη θα τα κατάφεραν καλύτερα εκτό Ευρωζώνης με ε, ανατιμημένο νόμισμα. Ευχαριστώ. Είχε το λόγο κυρία Αρκένα, αλλά δεν τη βλέπω εδώ. Δεν ξέρω, δεν παρίσταται. Το λόγο έχει ο κύριος Λούχαν. κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι ουσιώδες κατά τις συζητήσει για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη 24 η και 25 η Μαρτίου να έχουμε ένα μια αξιόπιστη δέσμη νομοθετικών μέτρων όσον αφορά την παγίωση τη οικονομική διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτική συνοχή, καθώς και η κοινή γεωργική πολιτική είναι δύο πυλώνες για το νέο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ουσιώδες η πολιτική συνοχής να διατηρήσει το μέρος που της ανήκει ε, στον ε, μελλοντικό προπολογισμό, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να εκπληρώσει του φιλόδοξου ε, στόχου του και να υλοποιήσει του στόχους της Ευρώπη 2020. Η πολιτική συνοχή πρέπει να οδηγήσει σε επενδύσει με στρατηγικά προγράμματα επενδύσεων, να επικεντρωθεί σε στόχου κλειδί κλπ. Έχει το λόγο ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα αντιμετωπίσουμε θέματα που αφορούν την τροποποίηση της ε, συνθήκης Λισαβόνας σε ό,τι αφορά το μηχανισμό σταθεροποίησης για τα οικονομικά θέματα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση και αυτό μας υποχρεώνει να έχουμε μια καλύτερη μορφή συντονισμού των οικονομικών μέτρων. Και αυτός ο μηχανισμός αφορά την ε, ζώνη του ευρώ. Βέβαια, οι χώρες οι οποίες είναι εκτός της ζώνης του ευρώ δεν θα επηρεαστούν από, τον, από τις αλλαγές αυτές. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διατηρήσουμε την ε, γενική ισχύ των κανόνων και θα πρέπει να υπάρξει και μία αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην θεωρούμε ότι μόνο οι χώρες του ευρώ βρισκόνται σε μία κλειστή λέσχη. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρχει μια απόλυτη ισότητα όλων των χωρών σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η κυρία Μπένοβα, Φασίκοβα Μπένοβα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο πτυχές πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Λοιπόν, η δουλειά των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θα αποδυναμωθούν από τις αποφάσεις που ίσως ληφθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα εθνικά κοινοβούλια θα έχουν όλο και λιγότερο πεδίο και δυνατότητες για να επηρεάσουν διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής και θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι αντιπαραγωγικό. Πώς θα πετύχετε ανάπτυξη και απασχόληση από αυτά τα μέτρα. Αυτό ο συνδυασμό των μέτρων δεν θα βγάλει την Ευρώπη από την κρίση. Αντί από περιοριστικά και μη δημοκρατικά μέτρα και πολιτικέ, εγώ θα ήθελα, και εδώ διακόπτω το μικρόφωνο τη ομιλήτρια. Τελευταία κυρία Γιακονσάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Γιακοσάρη. Έχουμε, όπως ξέρετε, άσχημα νέα από την Πορτογαλία. οι συντηρητικοί έχουν ζητήσει νέες εκλογές ή το κόμμα της αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο μπορεί να έχει συνέπειες για τη σύνολη κρίση στην Ευρωζώνη. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει προφανώς αρνητικές ε, επιπτώσεις και οι αγορές θέλουν μια ταχεία λύση και μια αξιόπιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων στην Ευρωζώνη. Πρέπει να βρεθεί μια λύση και μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο το ζήτημα αυτό, διότι έχουμε και το ζήτημα του συντονισμού που έχει κεντρικό χαρακτήρα. Τα κράτη-μέλη μας πρέπει να δημιουργήσουν μια νέα αρχιτεκτονική για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή όλο αυτό το σχέδιο έχει το άρωμα του νέου φιλελευθερισμού και αυτό του δίνει μια λανθασμένη αρνητική, θέση. Κλείνουμε και δίνουμε τώρα το λόγο στον Επίτροπο Όλη Ρεν και για να απαντήσει εξ ονόματος της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου θέλω να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα υπεύθυνη αυτή συζήτηση που διενεργήσατε σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας και θα ήθελα εξ ονόματος της Κομισιόν να κάνω μια σειρά σχολείων για κάποιες παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων και κυρίω να αναφερθώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ιαπωνία πριν έρθω στα οικονομικά θέματα. Η Κομισιόν, όπω ξέρετε, δεν έχει κάποια αρμοδιότητα για θέματα ασφάλεια και άμυνας. Βέβαια, έχουμε προσπαθήσει να συντονίσουμε για την κατάσταση στη Λιβύη, λοιπόν, έχει γίνει μία εφαρμογή του ψηφίσματο 1973 των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα η ζώνη μη υπερπτήσεω, και όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να λάβουμε υπόψη μα όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική αρρωγή που θα πρέπει να δώσουμε σε όλου αυτού, οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτή τη βοήθεια, είτε στην Λιβύη είτε στα σύνορα τη Λιβύη. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα φυστούμε των ζώων των αθών. Για τα γεγονότα στην Ιαπωνία πάλι. Τα γεγονότα αυτά δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να καταγράψουμε τα ενδεχόμενα προβλήματα που υπάρχουν στις πυρηνικές πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που είναι στη διάθεσή τη για να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο στα θέματα Ασφάλεια των αντιδραστήρων και επίσης σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων. Μας δίδαξε βέβαια η Ιαπωνία ότι οι κίνδυνοι μπορούν κάποτε να πραγματοποιηθούν. Αλλά όλα αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και στη σωστή μας σχεδίαση. Να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών ώστε να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την προστασία που παρέχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. του φτάσω σε τελικά συμπεράσματα σε σχέση με το ατύχημα αυτό στην Ιαπωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την αξιολόγηση που θα καλύψει τα πιο σημαντικά θέματα όπως είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας σε περίπτωση σεισμών και επίσης και τις προδιαγραφές για να εξασφαλίζεται η ψήξη των αντιδραστήρων. Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική, νομίζω ότι η συζήτησή σας καταδεικνύει τα διακυβευόμενα στην αυριανή συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα οποία είπατε θα γίνουν ακουστά από όλους σε όλες τις πρωτεύουσε της Ευρώπης. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει εξελιχθεί σημαντικά μετά από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει γίνει η οικονομική κρίση ουσιαστικά μια κρίση πολύπλευρη και στον τραπεζικό τομέα και στον οικονομικό στίβο και αυτό υποχρέωσε την Ευρώπη να αναζητήσει νέες δυνατότητες να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις και να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα έχουν μακρόπνοες συνέπειες. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαρόσο στις εναρκτήριες του παρατηρήσεις, θα απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση με μια συνολική στρατηγική που βασίζεται στην ισχύ, στους θεσμούς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιου είδους προκλήσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι αυτές που είχε σαν στόχο να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε από κοινού να αντιμετωπίσουμε αυτές τις θύελες και με τις κοινέ μας προσπάθειες να εξέλθουμε από δύσκολες καταστάσεις ενισχυμένοι και ευρωστότεροι. Ως αποτέλεσμα λοιπόν διαπραγματεύσεων που χρειάστηκαν πολλούς μήνες έχουν αναδυθεί τώρα τα στοιχεία για μια συνολική αντιμετώπιση σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Έχουν συμφωνήσει σε αυτά οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένουμε να επικυρώσουν τα στοιχεία αυτά αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη και ιδίως τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ εξακολουθούν να καταβάλουν έντονες προσπάθειες για δημοσιονομική παγιοποίηση και προχωρούν με μεγάλη αποφασιστικότητα τις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό τους. Αυτό είναι και ο ακρογωνίας λίθος της προόδου για τα θέματα αυτά. Και κατά δεύτερο λόγο, τόσο το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο είναι προσιλωμένα στη δέσμευσή τους να εξασφαλίσουν ότι το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης θα έχει περατωθεί και διεκπερωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση γιατί αυτή είναι προϋπόθεση και αγκονάρι της απάντησης που δίνουμε στην κρίση. Ο μόνιμος μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων στην Ευρώπη θα λειτουργήσει από τον Ιούνιο του 2013 με ικανότητα δανειοδότησης πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτή την απόφαση εμείς θα έχουμε ένα σύστημα ασφαλείας στον χρηματοοικονομικό χώρο με αρκετή ικανότητα συγκράτησης ώστε να διαλύσει ακόμα και τις πιο ελάχιστες αμφιβολίες σε σχέση με την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει δυσμενή οικονομικά σενάρια. Ο ρόλος της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού θα είναι κεντρικός και η σύνδεση του μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμπεριλαμβάνουν προφανώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθοριστεί με μεγάλη σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Εν καιρό θα προτείνουμε και ένα κανονισμό ο οποίος θα βασίζεται στο άρθρο 136 <clears throat> της συνθήκης που θα διευκρινίζει τα βήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να εξασφαλίσουμε τις πολιτικές κατευθύνσεις και την συμβατότητα με τα πλαίσια παρακολούθησης των επιμέρους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταίο αλλά όχι και ίστατο είναι το θέμα ότι η μεταρρύθμιση του, χρήμα, του τραπεζικού πιστοτικού τομέα θα πρέπει να διαφυλαχθεί η σταθερότητά του για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν οι τράπεζες να δανείζουν στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες. Το επόμενο κύμα stress test των τραπεζών θα γίνει στους επόμενους μήνες και θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες αναδιάθρωσης και ενδεχομένω ανακεφαλοποίηση στον τομέα των τραπεζών. Προτού δημοσιευθούν τα αποτελέσματα, όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν ποιε θα είναι οι στρατηγικές τους και να τις παρουσιάσουν εάν αυτό καταστεί απαραίτητο για την αναδιάθρωση και επανακεφαλοποίηση τροτών τραπεζικών τους φορέων. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα επιληθούν εν παραλληλία. Χρειάζεται να εξασφαλιστεί με μεγαλύτερη ταχύτητα η αναδιάθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και ενδεχομένως επανακεφαλαιοποίηση αν αυτό είναι απαραίτητο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα γιατί αυτό πολύ μια προϋπόθεση για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία και να διατηρηθεί η σταθερότητα και το εύρωστο των τραπεζών και η εξασφάλιση και η διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από την παροχή πιστώσεων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει την δεσμευσή του για την υλοποίηση όλων αυτών των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην συνολική μας οικονομική στρατηγική για την υπέρβαση της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να αναστρέψει το, ε, την τάση στο εφετινό οικονομικό έτος. Αυτό δεν σημαίνει το τέλος της κρίσης, ούτε ότι μπορούμε να επαναπαυόμαστε. Σημαίνει όμως ότι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις και για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους κρίσεις στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το λόγο για το Συμβούλιο ο Υπουργός Γιώρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευγνωμονώ ιδιαίτερα για αυτούς που πήραν μέρος στη συζήτηση και οι περισσότεροι αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ανάγκη για τα έξι στοιχεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση και να δώσουμε μια κοινή απάντηση ως Ένωση. Και ελπίζουμε οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων την Πέμπτη να το αποφασίσουν αυτό και να βάλουμε τις βάσεις για την πρόληψη παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον. Επίσης συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι δεν περνάει η Ένωση, Ένωση κρίση, αλλά κράτη-μέλη τα οποία μπλέχτηκαν μέσα σε, μια, σε ένα σπυροειδές χρέωσης. Και αυτός είναι και ο κύριος στόχος αλλά όλοι μας είμαστε μέλη μιας ένωσης. Έχουμε κοινή νομισματική πολιτική, έχουμε κοινό νόμισμα. Η κρίση λοιπόν μιας χώρας πρέπει να τη μοιραστούμε όλοι, γι' αυτό χρειαζόμαστε κοινή απάντηση. Ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα πρέπει να την διαχειριστούμε για διαπραγματεύσεις για τα έξι αυτά νομοθετήματα όσον αφορά την ε, διακυβέρνηση, τη διάκριση μεταξύ καλών και κακών πιστώσεων. Αν υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και η Κομισιόν θα σας το επιβεβαιώσει ότι συζητήθηκε αυτό στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο έχει ορισμένους δισταγμούς σχετικά με, τις, με, το καλό χρέος, με το καλό Γιατί πολλές φορές το καλό χρέος φαίνεται καλό και μετά αποδεικνύεται διαχρονικά ότι είναι ένα αρνητικό φαινόμενο. Συζητιέται λοιπόν το θέμα αυτό, διότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση πρέπει να ενθαρρύνουμε την οικονομία, να κινητοποιήσουμε την οικονομική ανάπτυξη με άλλους τρόπους και όχι μόνο χρησιμοποιώντας χρέος. Δεν θα πρέπει να χρεώσουμε τις μελλοντικέ γενιές. Πρέπει να κάνουμε καλές επενδύσεις σήμερα, όχι σε βάρος των επόμενων γενιών. Γι' αυτό πολύ σωστά είπε ο κύριος Μπαρόσο, πρέπει να έχουμε τα σωστά μέσα στα χέρια μας, να ενισχυθεί περισσότερο η, η ενιαία αγορά, να αρθούν τα εμπόδια που υπάρχουν κλπ. Τώρα δύο λόγια για την κατάσταση στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Για την Πορτογαλία στις 11 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων επικρότησαν το πορτογαλικό πακέτο το οποίο τότε ανακοινώθηκε και η Κεντρική Τράπεζα επίσης το επικρότησε ήταν ένα θετικό μήνυμα για τις αγορές αυτό, Όμως οποιοδήποτε πρόγραμμα αξίζει μόνο αν εφαρμοστεί. Θα πρέπει να υπάρχει πολιτική δέσμευση για κάθε πρόγραμμα, ειδικά για την Ιρλανδία δε, έχω να πω ότι η νέα κυβέρνηση έδειξε πνεύμα συνεργασίας στο Γενικό Συμβούλιο και ελπίζω στη συνάντηση του Συμβουλίου να είναι σε θέση να βρεθούν οι σωστές απαντήσεις στην Ιρλανδική κρίση με από κοινού με της Ιρλανδικής κυβέρνησης. Κοινοτική μέθοδος ή διακυβερνητική μέθοδος. Συχνά τίθεται αυτό το ερώτημα. Από τις 4 Φεβρουαρίου έχουμε διανύσει μεγάλο δρόμο. Στις 4 Φεβρουαρίου πολλά από τα κράτη-μέλη και πολλοί ευρωβουλευτές φοβόντουσαν για το τι θα συμβεί αν σημαντικά θέματα φεύγανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ξαναγυρίσαμε στο μεταξύ στην κοινοτική μέθοδο και αυτό βελτίωσε την κατάσταση και ως Προεδρία έργο μας είναι να πείσουμε όλους να βρεθεί συνένεση. Μερικοί αυτών που θέλουν να αφαιρεθούν ορισμένε αρμοδιότητε από την Ένωση και των υπολείπων. Ο Πρωθυπουργό τη Ουγγαρία ήδη στι 4 Φεβρουαρίου είπε ότι στα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πρέπει να γίνεται μνήμα του, του ότι ε, δρούμε με βάση τη συνθήκη. Το ίδιο και για το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας όπως ονομάζεται τότε. Και για να ξαναγυρίσω, ξαναγυρίσω μάλλον στην κοινοτική μέθοδο στο μεταξύ και η Κομισιόν που είναι το πιο το, το πραγματικά κοινοτικό όργανο επιφορτίστηκε Επίσης εγγύησεις δόθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρόσβαση στις πληροφορίες. Νομίζω κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Το, ε, το σύμφωνο για το ευρώ είναι και αυτό μια νέα δημιουργία. Οι χώρες μέλη όπως η Ουγγαρία, αν θέλουν, μπορούν να μπουν στο ευρώ, παρότι ακόμα δεν έχουμε το ευρώ ως νόμισμα. Και τέλος, επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για την πιο επικοδημητική προσέγγιση σε σχέση με τη συζήτηση που θα γίνει για το πακέτο αυτό για την οικονομική διακυβέρνηση. Οι εκθέσεις των Ευρωβουλευτών που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο ελήφθησαν υπόψη στην ε, διαμόρφωση των πορισμάτων του Συμβουλίου. Λιβύη και Μεσόγειος. Πόλεμος και αστάθεια είναι οι πιο μεγάλες κρίσεις για αυτούς που ζουν στην περιοχή αυτή, αλλά είναι απειλή και για την Ευρώπη, όπως ε, είπε ο κύριος Μάουρο και συμφωνώ. Επίσης είχαμε την ευκαιρία και αυτό να το μετατρέψουμε σε θετική εξέλιξη και να αποτρέψουμε περαιτέρω τραγωδία στην περιοχή, στη Μεσόγειο. Είμαι υπέρ του, της ειλικρινούς ομιλίας και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο αντέδρασε πιο γρήγορα από ότι το Συμβούλιο στο θέμα αυτό. Την τελευταία στιγμή μόνο καταφέραμε να κινήσουμε μια δράση με τον συνασπισμό παρεμβαίνοντας στη Βεγγάζη και αυτό έσωσε τις ζωές πολλών. Τώρα, σε τι βαθμό, στο βαθμό μάλλον που είμαστε ενωμένοι και στο βαθμό που κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας για την Ένωση είναι αποτελεσματική, αυτό πρέπει να το συζητάμε με ειλικρίνεια, διότι δεν είμαστε ενωμένοι 100%. Πολλά θέματα βέβαια συμφωνούνται πρέπει να βρεθεί η σωστή απάντηση και αυτό είναι θετικό. Στις 11 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι Πρωθυπουργοί δήλωσαν ότι ο Καντάφη πρέπει να φύγει και ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί επαφή με το Λιβικό Συμβούλιο και οι Λιβικές Αρχές θα πρέπει να ζητήσουν βοήθεια για τη χώρα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με τους νότιους γείτονες, δεδομένου ότι έχουν αρχίσει δημοκρατικές αλλαγές και πρέπει να τις βοηθήσουμε. Χρειάζεται οικονομική βοήθεια, υπό όρους βέβαια. Πρέπει να στενέψουν οι οικονομικοί δεσμοί, να βοηθήσουμε τις κοινωνικές αλλαγές στην περιοχή με βάση τους τρεις στόχους πρόσφαση στην αγορά, κινητικότητα και το οικονομικό. Στις 21 ε, Μαρτίου οι Υπουργοί Εξωτερικών επανέλαβαν αυτές τις δεσμεύσεις. Στο μεταξύ το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε πάρει την απόφαση 1973 την οποία επικρατήσαμε όπως επίσης και η απόφαση της διάσκεψης του Παρισιού και η εφαρμογή ξεκίνησε. Δράσαμε γρήγορα όσον αφορά τις κυρώσεις και επαναλάβαμε την δέσμευσή μας να βοηθήσουμε τον άμαχο πληθυσμό στη Λιβύη. Η κοινή εξωτερική πολιτική μπορεί να μην είναι αποτελεσματική στη δράση της, πάντως, έστω και την τελευταία στιγμή, εγκαίρως τουλάχιστον, ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Περατώθηκε αυτή η συζήτηση. Και τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε την δήλωση του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την κατάσταση στην Ιαπωνία, όπως επίσης και τον συναγερμό στους πυρηνικούς σταθμούς.